Bene. Come si fa qua? Vabbè, non sono capace. E prego, colleghi, se volete accomodarvi, direi di cominciare anche perché abbiamo eh, un'importante. Καλή σας ημέρα. Αν θέλετε α ξεκινήσουμε γιατί έχουμε σημαντικέ ψηφοφορίε. Έχω να σα κάνω και κάποιε ανακοινώσει και στι 10 θα έρθει η Υπουργό παιδεια τη Ιταλία. η Στεφάνια Τζανίνη να μα παρουσιάσει τι προτεραιότητε τη Ιταλική Προεδρία σε αυτό το τομέα. Ξεκινάμε το σημείο 6 τη ημερησία διάταξη. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Δεν ξέρω αν είχατε χρόνο να διαβάσετε αυτές τις αποφάσεις. Ε, είναι διαθέσιμες από αργά χτες μόλις ε, λυπάμαι γι' αυτό ε, να σας τις ε, υπενθυμίσω εντάχει έτσι ώστε να είστε ενήμεροι και ενήμερες σημαντικές αποφάσεις πρώτη απόφαση κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος της θητείας μας θα διατηρήσουμε το σύστημα των πόντων για την ανάθεση εκθέσεων. Είναι το σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί η Επιτροπή μας από το 1999 και μετά. Δεύτερον, στο μέσον της ε, κοινοβουλευτικής μας θητείας θα αναθεωρηθεί το σύστημα. Τώρα, χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων προβλέπει πολλά απογεύματα πέμπτης. Όχι μόνο για τη δική μας επιτροπή, αλλά και για άλλες. Ε, για λόγους ε, οργανωτικούς και πρακτικούς η γραμματεία ανέφερε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μειωθεί ο αριθμός των απογευμάτων πέμπτης που θα πρέπει να συνεδριάσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι η πέμπτη είναι μια μέρα δύσκολη. Άλλη απόφαση. Θα πρέπει μαζί με τους συντονιστές να συντάξουμε εκ των προτέρων τις γραπτός τις τρεις ερωτήσεις που έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε στον υποψήφιο ε, Επίτροπο. Όλοι οι ευρωβουλευτές από την άλλη μεριά έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της ακρόασης να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν. Οι συντονιστές θα υποβάλουν τις ερωτήσεις των ε, ομάδων μόνο. Άλλο θέμα. Οι συντονιστές ζήτησαν από την Πρόεδρο να στείλω ε, επιστολή στον πρόεδρο τη Επιτροπή των Περιπολογισμών με στόχο να διευκρινιστεί η θέση της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά την τροπολογία του συμπληρωματικού ε, τροποποιητικού προπολογισμού του 2014. Ε, το πρόβλημα αφορά τις πληρωμές του 2014. Το Συμβούλιο ε, αποφάσισε να επανακτήσει τα ποσά τα οποία έλειπαν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει πριν το τέλος του 2014 που θα εγκριθούν τα πολυετή προγράμματα. Όμω αυτό δεν έχει γίνει, δεν ούτε πρόκειται να γίνει τελικά. Το υπενθυμίσαμε στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου χτες. Σήμερα θα το υπενθυμίσουμε και στην Υπουργό. Γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση το 2014 και αυτό είναι το Εράσμους. Καταλαβαίνετε τι συνέπειε μπορεί να έχει αυτό. Οι συντονιστέ αποφάσισαν επίση η Επιτροπή πολιτισμού να ζητήσει την άδεια να προβεί στη σύνταξη δύο εκθέσεων ε, πρωτοβουλίας, ιδίας πρωτοβουλίας. Μία σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Κομισιόν για την συνολική αντιμετώπιση πολιτικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η ομάδα των φιλελευθέρων με δύο πόντους θα έχει έναν εισηγητή και το ΕΛΚ ένα εισηγητή με τους δικούς του πόντους για μια έκθεση περί της ανακοίνωσης κομισιών για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες στην ψηφιακή εποχή. Θα προσπαθήσουμε επίσης να δούμε ποια είναι η κατάσταση με το Ευρωπαϊκό ε, ε, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Ε, σκεφτόμαστε να οργανώσουμε ένα σεμινάριο με τους υπεύθυνους αρχιοθέτησης της, στη Φλωρεντία. Τι έγινε τώρα με την, τον προπολογισμό για την έρευνα του 2014. Σας εξηγήσω. Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο του, ε, της, του Τμήματος Πολιτικής ε, που προβαίνει σε μελέτες και μετά την Υπουργό θα ακούσουμε ε, τις εργασίες του ε, τμήματος αυτού για την ε, έκθεση περί διπτής εκπαίδευσης. Θα πρέπει όμως να δούμε αν οι τέσσερις εκθέσεις που είχαμε προβλέψει μπορούν να εγκριθούν για να μην χάσουμε τα ποσά του 2014. Θα πρέπει να μας πείτε όμως αν συμφωνείτε με αυτές τις τέσσερις μελέτες τις οποίες είχαμε προαποφασίσει. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα για να αποφασίσουμε, αλλά ε, ο χρόνος πιέζει. Το πρόγραμμα του 2015 βρίσκεται ήδη στα χέρια της Κομισιόν. Επίση, θα πρέπει να αποφασίσουμε για το κατά πόσο να χρησιμοποιήσουμε τι ε, δημόσιε ακροάσει προ την Κομισιόν, με την Κομισιόν. Ε, έχουμε την ημερομηνία της 22 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δώσουμε απαντήσει σε αυτά τα θέματα και να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που εκκρεμούν. Και μετά έχουμε και κάποια πιο πολιτική απόφαση. Ε, οι συντονιστές αποφάσισαν να σταλεί επιστολή στον πρόεδρο Γιούνκερ για να υπογραμμιστεί η σημασία του χαρτοφυλακίου του, της παιδείας και, της, του πολιτισμού έτσι ώστε ο αντίστοιχος επίτροπος ε, να έχει μια πιο σφαιρική προσέγγιση να γνωρίζει τα θέματα της ψηφιακής εποχής και των ε, προϊόντων του διαδικτύου. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι θέλουμε ίση μεταχείριση, διότι πιστεύουμε πως ο πολιτισμός μπορεί να οθήσει την ανάπτυξη της Ευρώπης τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτά. Ας περάσουμε στις πληροφορίε για τον προϋπολογισμό του 2015. Έχετε τις κάρτες σας, φαντάζομαι έτσι δεν είναι. Βάλτε τις στην αντίστοιχη σχισμή. Σημεία 7 και 8 της ημερησίας διάταξης λοιπόν. Έχουμε δύο κατάλογοι ψηφοφοριών διαφορετικοί. Ένας κατάλογος για τους αριθμούς, για τα νούμερα και ένας άλλος για, με τις ε, προτάσεις του εισηγητή. των, της συγγήτρια συγκεκριμένα. Έχουμε τα προγράμματα Marie Εράσμους Erasmus κλπ. Ε, τα οποία πιστεύουμε πως ε, πρέπει να ε, πάρουν περισσότερη χρηματοδότηση. Θέλουμε να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε το 2015. Οι περικοπές που έγιναν στο, στο ε, ε στο Marie Κιουρί κλπ. δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερη χρηματοδότηση, πιο πολλά κονδύλια από το Συμβούλιο, να το ξανασκεφτεί, γιατί οι περικοπές 3,5% είναι απαράδεκτες. Γιατί, γιατί θα θέσουν σε κίνδυνο την ορθή υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Είπαμε ότι θα στείλουμε και την επιστολή αυτή στην Επιτροπή Προπολογισμών, την οποία αποφάσισαν οι συντονιστέ. Γιατί θέλουμε ότι το 2015 το Εράσμος να έχει επαρκή κονδύλια. Ε, το πρόβλημα των πληρωμών οριζόντιο επηρεάζει και άλλες επιτροπές, άλλα προγράμματα επίσης του Κοινού ε, άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο για τα δημοσιονομικά θα προσπαθήσει να βρει μια λύση σε αυτά τα οριζόντια θέματα συνολικά. Περνάμε στο σημείο 7. Κατάλογος ψηφοφοριών, όπως σας είπα, το έχει όλες τα νούμερα. Οι και είχαμε και μια προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 23 Ιουλίου, 26 τροπολογίες κατατέσκαν και συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τις ομάδες και τους κοιόδης εισηγητές και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που κατάφεραν να βρουν μία όσο το δυνατόν περισσότερο συνενετική λύση. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1. Ε, υπέρ. Α, ένα λεπτό. Ε, ένα λεπτό λέει η πρόεδρος. Ε, είχα το λάθος έγγραφο στα χέρια μου. Α, τροπολογία 24. Κβάντα Μίτσι Μοργάνο Αγοράκης υπέρ διανατάσεως της χειρός παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 5703 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 5704. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 05. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, η 6. Συμβιβαστική τροπολογία 1 Συμβιβαστική 1. Σελίδα 3. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. προπολογια τροπολογία, 57-08 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Πιο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική στην τροπολογία 2. Ε, αφορά δύο τροπολογίες. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Μαλτέζε κλπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 έχει αποσυρθεί. Ε, συμβαστική πρόταση παριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην τροπολογία, σημαντική τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, Jill Evans και πάλι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, διακόνου κλπ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, βέντα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαρθμών 20, παραντίκα και άλλων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 καβαντά και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 καβαντά και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στον, στο δεύτερο κατάλογο ψηφοφοριών. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση, τροπολογία υπαριθμών 1 τρούπελ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Όχι, όχι, όχι, πάμε κατευθείαν στην 3. Ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμών 4. Λιμπάτσκα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 5. Νιριάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ε, πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την, ε, το Συμβούλιο Υπουργών, μετά την συνεδρία του, του, του Συμβουλίου Υπουργών. Ε, προφορική τροπολογία λοιπόν. Έλγα Τρίπελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 7. Έχουμε μια χωριστή ψηφοφορία εδώ. Ε, με αίτημα των σοσιαλιστών. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία παριθμών 2, ε, υπέρ, κατά, αποχές, συγγνώμη ξανά, υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονική ψηφοφορία για επιβεβαίωση γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Allora, ah, scusate, eh, ah, ehm, considero aperta la... Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα 23 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Οπότε απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. Τροπολογή παριθμών 1. Io ho letto Συγγνώμη, το διάβασα λάθος εγώ. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Εγώ έκανα λάθο, λέει πρόεδρο. Ε, τροπολογία Ε, συγγνώμη, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. τροπολογία υπαριθμών 12 υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 13 του εισηγητή και πάλι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, προφορική τροπολογία υπαριθμών 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 15, λιμπάτσκα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 4, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, Νιριάντα, όχι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι, 17. 17. Νιριάντα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η 18, πάλι Νιριάντα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα πρέπει να κάνουμε την, να δώσουμε την τελική μας γνώμη για το σύνολο του σχεδίου της νομοδότησης. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Κλείνει η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα... Allora, allora, pur 24 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά, 0 αποχές. 24 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε μαζί. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη μάχη στην Επιτροπή Προπολογισμών και γενικότερα με όλο το Κοινοβούλιο ε, πρέπει να προσπιστούμε αυτών των αυξήσεων που ζητάμε και να δώσουμε ένα πραγματικό μήνυμα ε, κατά των περικοπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και πάλι. Μπορούμε τώρα να διακόψουμε την συνεδρίαση μέχρι τις 10 όταν θα έρθει ο υπουργό. Θα είναι κοντά μας. Λοιπόν, 20 λεπτά διακοπή μέχρι τις 10 η ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Αν έχετε την καλοσύνη, διακόψτε τις προσωπικές συζητήσεις. Και θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση που έχουμε μαζί μας σήμερα την Υπουργό Παιδείας από την Ιταλία. Η ε, κυρία Στεφανία Τζανίνη. Λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την έχουμε μαζί μας σήμερα. Πρόσφατα είχε μια σημαντική ακρόαση με την Επιτροπή Ήτρε για την έρευνα και σήμερα θα μας μιλήσει για την παιδεία και τα πανεπιστήμια. Στεφανία, σε ευχαριστώ που ήλθες. Ε, έχουμε δε αυτή τη συζήτηση σήμερα αντί για χθες που συναντηθήκαμε με τους άλλους υπουργούς γιατί υπήρχε μια σημαντική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ιταλία χθες για τη μεταρρύθμιση των σχολείων. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που ξαναγύρισες στις Βρυξέλλες σήμερα για να μας δεις. Ήσουν εδώ πριν από λίγες μέρες. Έλεγα λοιπόν ότι θέλουμε πολύ να ακούσουμε για όλα τα θέματα ε, που συζητούσαμε στην τελευταία θητεία του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, το, το Συμβούλιο ε, ε, έκανε περικοπές στα προγράμματά μας, σε κάποια από τα προγράμματά μας. Και θα θέλαμε σήμερα να δούμε αν έχουμε κάποια θετικά μηνύματα για την επαναφορά αυτών των κονδυλίων για το 2020, το πρόγραμμα Εράσμους κτλ. Είναι προγράμματα που είναι σημαντικά, αλλά έχουν υπάρξει περικοπές για το 2015. Θέλουμε λοιπόν η Ιταλική Προεδρία και εσύ προσωπικά να κάνεις κάτι για να ανατρέψεις αυτές τις περικοπές. Ε, μόλις ανασκοπήσαμε τον προϋπολογισμό σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας και υπήρχε, υπήρξε ευρεία συνένεση να επιμείνουμε στην επαναφορά. Στην επαναφορά των κονδυλίων που μας αφαιρέσανε για τα προγράμματα, από τα μας. Το 2015 ευτυχώς το Εράσμους ε, έχει περισσότερα κονδύλια καθώς και πιστώσεις πληρωμών. Όμως στην, στον τροποποιημένο προϋπολογισμό για το 2014 οι πληρωμές για το Εράσμος δεν έχουν αποκατασταθεί και ανησυχούμε γι' αυτό διότι αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις και για το μελλοντικό πρόγραμμα. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε εκατομμύρια από νέους Ευρωπαίους. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια ε, φοιτητές που ενδεχομένως θα συμμετάσχουν ε, θα είναι απογοητευτικό να μην έχουν κονδύλια το πρώτο έτος της επόμενης περίοδου. Σας σε παρακαλούμε λοιπόν να επιμείνεις για την αποκατάσταση των κονδυλίων. Τώρα λοιπόν θα σου δώσω το λόγο και βεβαίως μετά θα υπάρξουν και ερωτήσεις από συναδέλφους. Ευχαριστώ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβια. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, καλημέρα. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση να είμαι μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, η συνάντηση αυτή είχε προβλεφθεί πριν από λίγες μέρες. Αναφέρθηκε σε αυτό η Πρόεδρος. Όσον αφορά τη στρατηγική προσέγγιση ε, της παιδείας στην Ιταλία υπήρχε αυτή η σημαντική συνεδρίαση χθες. Σήμερα χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για τις σκέψεις της Ιταλικής Προεδρίας για την παιδεία. Η Ιταλική Προεδρία βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση, πρέπει να σας πω, για διάφορους λόγους. Ο πρώτος από αυτούς είναι ότι η Προεδρία μας συμπίπτει με την εκκίνηση του νέου ε, προγραμματισμού, επταετούς προγραμματισμού των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Έχουμε και τον ορίζοντα του 2020 και το Erasmus ε, Δεν αφορά μόνο την κινητικότητα των φοιτητών πανεπιστημίων. Είναι ένα φιλόδοξο και στρατηγικό πρόγραμμα το Erasmus Plus για την αμοιβαία αναγνώριση για τη δημιουργία του χώρου των γνώσεων στην Ευρώπη. Συνεπώς, έχουμε ε, σοβαρές ευθύνες να διεκπαιρεώσουμε και πρέπει να υποβάλουμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα. Αν περάσουν αυτές οι αυτοί οι προσανατολισμοί μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλαίσιο αναφορά στον νέο ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες όταν θα σας μιλήσω για τις δραστηριότητες. Μία άλλη σημαντική περίσταση ε, που αντιμετωπίζουμε είναι πολιτικής φύσης. Η Ιταλία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της μεταβατικής περίοδου από την παλιά Κομισιόν στη νέα. Και ε, έχουμε και ένα νεοεκλεγέν Ευρωκοινοβούλιο. Συνεπώς αυτή η Προεδρία, η Ιταλική, ε, πρέπει να μπορέσει να σπείρει σωστά τους σπόρους που θα αποδώσουν τους καρπούς επόμενες, τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς έχουμε αναπόφευκτες ευθύνες, Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, είμαστε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας στο Ευρωκοινοβούλιο, με σας. Έχουμε τέσσερις μήνες μπροστά μας και μέχρι το τέλος θα δουλεύουμε μαζί εντατικά και ελπίζω ότι θα έχουμε κοινέ προτεραιότητες για τον προγραμματισμό. Γενικά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες μας. Ε, ας πάρουμε τα προγράμματα και τις ανάγκες. Τις ανάγκες ανασκόπησης, αν θέλετε, αναθεώρησης της ατζέντα για την παιδεία και την κατάρτιση στην Ευρώπη. Το πλαίσιο της κρίσης είναι διαρθρωτικό ενδεχομένως περισσότερο παρά κυκλικό. Δηλαδή, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση μόνο ε, πετύχουμε σημαντικές επενδύσεις και από την άποψη την χρηματοοικονομική αλλά και από την άποψη την πολιτιστική. Δηλαδή χρειαζόμαστε και ιδέες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τις δομές της παιδείας και της έρευνας. Την παιδεία τη χρειαζόμαστε διότι θέλουμε να έχουμε όλο και περισσότερο γνώση στην Ευρώπη του αύριο. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ακόμη ότι οι νέοι μας θα έχουν όλο και περισσότερο τις ε, συγκεκριμένες ικανότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τη σταδιοδρομία τους. Έχουν πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση για αύριο. Και υπάρχει και η έρευνα μίλησα για την έρευνα σε άλλη επιτροπή, αλλά θέλω να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να επιστρέψει στην ανταγωνιστικότητα. Έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκή ατζέντα για αυτά τα τρία θέματα. Η ατζέντα αυτή προβλέπει τη συνεργασία ώστε να συμμετέχει περισσότερο η κοινωνία, να υπάρχει αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει συνεπώς να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Η βάση του Ιταλικού προγράμματος, όπως έχετε υπόψη σας, σίγουρα είναι η εξασφάλιση της ανάπτυξης της απασχόλησης, της την οποία θέλουμε να προωθήσουμε και αριθμητικά και ποιοτικά και ακόμη θέλουμε να έχουμε ένα χώρο ασφάλειας και ελευθερίας ώστε πραγματικά να μπορούν οι άνθρωποι να χαίρουν των δικαιωμάτων τους και να παίξει και η Ευρώπη ένα πιο στρατηγικό ρόλο στον κόσμο. Η Προεδρία λοιπόν θα ακολουθήσει αυτές τις τρεις κατευθυντέριες γραμμές όταν εξετάζει την ευρωπαϊκή πολιτική. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές που έχουμε εντοπίσει θα ενισχύσουν το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Βασική μας προτεραιότητα είναι να εξετάσουμε σε βάθος το μελλοντικό ρόλο της παιδείας σε σχέση με την ανάπτυξη αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην απασχόληση των νέων, την τεχνολογική προώθηση και την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων. Διότι δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν ε, εργασία με δεξιότητες παρά μόνο να αποκτήσουν τις δεξιότητες πριν. Ακόμη, εξετάζουμε και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, παιδείας μάλλον, και απασχόλησης. Στο Συμβούλιο της 12 η Σεπτεμβρίου έχουμε προτείνει να επικεντρωθούμε στην πολιτική συζήτηση του ρόλου της παιδείας ε, και της κατάρτισης μέσα στο πλαίσιο, στον ορίζοντα 2020 είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί αυτή η στρατηγική ώστε να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε αν θέλετε τους στόχους τους οποίους έχουμε ορίσει πριν από μερικά χρόνια ώστε να γίνουν υλοποιήσιμοι μελλοντικά. Θα ήθελα ακόμη να υπογραμμίσω την θετική ενέργεια, επίδραση των επενδύσεων στην παιδεία ώστε να εξασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων. Η ανεργία, το ξέρετε όλοι, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα στην Ευρώπη σήμερα. Θα έλεγα ότι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση ε, του ευρωπαϊκού συστήματος τριτογενούς κατάρτισης πρέπει να επανεξεταστεί. Δηλαδή, πρέπει να, κάνουμε, επιτύχουμε μια καλύτερη διαφοροποίηση των διαφόρων διαδρομών που προσφέρονται. Αυτό θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Και αυτό ισχύει για το πρόγραμμα των μαθημάτων και για το βαθμό ε, δέσμευσης μέσα στο πλαίσιο της παιδείας και αναφέρομαι στην πανεπιστημιακή παιδεία των παιδιών πάνω, άνω των 18 και χρειάζεται να έχουμε επαγγελματική κατάρτιση σαν στοιχείο το οποίο να εντάσσεται μέσα στις ακαδημαϊκές σπουδές και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα ε, επιστροφής στον... στην εκπαιδευτική διαδρομή ε, και στην κατάρτιση επίσης, επαγγελματική κατάρτιση είναι προφανές ότι χρειάζονται νέες δεξιότητες. Υπάρχουν εξελίξεις κάθε δεκαετία ε, και στις επιστήμες και στον τεχνικό χώρο και γι' αυτό είναι πολύ απαραίτητο οι άνθρωποι να μπορούν να ανανεώνουν τις γνώσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έχουμε και την αηφόρο ε, μάθηση. Παιδεία λοιπόν και ανάπτυξη. Αυτό δίνει και οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά ουσιαστικά εξασφαλίζει την ανάπτυξη για τους υπηκόους μας που θα μπορέσουν να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους μέσα στην οικονομική δυναμική της κάθε χώρας. Ένας από τους πιο καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης αυτής της διασύνδεσης μεταξύ παιδείας και ανάπτυξης θα αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου. Εκεί η Προεδρία θα υποβάλει τα συμπεράσματα όσον αφορά την παιδεία για την επιχειρηματικότητα. Μία από τις νέες ευρωπαϊκές ιδέες, αν θέλετε, είναι αυτή, αν και έχει αναγνωριστεί σαν σημαντικός παράγον σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά είναι κάτι καινούριο για τον ευρωπαϊκό χώρο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η διασύνδεση πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα συμπεράσματά μας θα προσδιορίσουν πώς καλύτερα μπορούμε να σμιλεύσουμε ένα επιχειρηματικό πνεύμα ενώ οι άνθρωποι είναι ακόμη μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιχειρηματικότητα ε, προσδιορίστηκε το 2006 στις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η ιδέα τότε ήταν να δώσουμε περισσότερες δεξιότητες σε όλους τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία συγκεκριμένη σπουδή, είναι μία διεπιστημονική προσέγγιση να προωθήσουμε την επινόηση, τη δημιουργικότητα, την ομαδική εργασία, την επίλυση ε, προβλημάτων. Και θέλουμε ακόμη να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους ε, να αναλαμβάνουν κινδύνους. Αυτό είναι ένα κομμάτι σημαντικό των φιλοδοξιών μας ε, και κάνουμε ένα βήμα μπρος σε σχέση με την ε, Ευρώπη ε, των παρελθόντων ετών. Είναι διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζομαστε μία μεταβολή της νοοτροπίας. Χρειαζόμαστε μία μετατόπιση του υποδείγματος αν θέλετε, του βέλτιστου δείγματος. Ε, πολλά πράγματα κινδυνεύουν ε, και οι άνθρωποι γίνονται λίγο πιο διστακτικοί στη διαχείριση των σταδιοδρομιών τους και ανησυχούν και για την αποτυχία προφανώς. Σε αυτή τη διαδικασία της πολιτισμικής ε, μετατόπισης, μετατόπισης νοοτροπίας πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες στάσεις ζωής και πρέπει να προετοιμάσουμε σωστά τους ανθρώπους για τον μελλοντικό κόσμο. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρώτα απ' όλα πρέπει να ε, καταρτιστεί σωστά ώστε να περάσει αυτή τη νέα νοοτροπία στους φοιτητές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ του χώρου των σπουδών και του χώρου της εργασίας είναι απαραίτητη. Χρειαζόμαστε και νέες διαδρομές για το εκπαιδευτικό μας προσωπικό. Είναι σημαντικό αυτό σαν προσέγγιση. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που στο Συμβούλιο των Υπουργών το Ευρωπαϊκό ε, έχουμε προβλέψει μια κοινή υπουργική συνάντηση Δηλαδή, ε, οι Υπουργοί Απασχόλησης θα προσκληθούν στους Υπουργούς Απασχόλησης και το αντίθετο θα συμβεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Ακόμη, θέλουμε να εξετάσουμε και το ρόλο της παιδείας στην ψηφιακή εποχή. 11 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί αυτό το θέμα στις Βρυξέλλες, συνεργαζόμαστε με την Κομισιό, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλουμε να δουλέψουμε στενά με την Επιτροπή σας πάνω σε αυτό, ώστε να ενισχύσουμε τις γνώσεις του ψηφιακού δυναμικού ε, και να εξασφαλίσουμε πρόοδο όσον αφορά το άνοιγμα των σπουδών της παιδείας. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αυτή. Ακόμη θα εξετάσουμε και την, το ρόλο της παιδείας στη μεταφορά αξιών. Και αυτό σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε μόνο μια ψηφιακή υποδομή θέλουμε να φροντίσουμε οι άνθρωποι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεχνολογία και πρακτικά και σε σχέση με τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε μια καλοριζωμένη μεταβολή των γνώσεων και του τρόπου που μοιράζονται οι γνώσεις. Θέλουμε νέες πρακτικές ε, διδαχής και θέλουμε ενίσχυση των γνώσεων. Νομίζω ότι αυτή η προτεραιότητα θα είναι κοινή και όλα αυτά, ιδανικά τουλάχιστον, θα αποτελέσουν ένα κοινό περιβάλλον παιδείας της Ευρώπης που θα ανανεώνεται συνεχώς, θα αναζωογονείται συνεχώς. Έχουμε και μία τρίτη προτεραιότητα που εντάσσεται στις προηγούμενες. Η σημαία της Ευρώπης σήμερα πρέπει να δώσει πιο σημαντική θέση στο Εράσμους. Έχουμε το Εράσμους Plus λοιπόν πρόγραμμα τώρα. Ε, αντιλαμβάνομαι την έκκληση που έκανε η Προεδρία να διατηρηθεί αυτός ο πυλώνας για τα επόμενα 7 χρόνια. Αλλά θέλουμε το Erasmus Plus να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για την διεθνή συνεργασία μεταξύ ανωτάτων ιδρυμάτων, ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα κινητικότητας μαζί με προγράμματα σπουδών. Συνεπώς και ε, ο στόχος μας είναι όμοιος με το Ευρωκοινοβούλιο και συνεργαζόμενοι φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε. Ίσως ξέρετε καλύτερα από άλλους, σε άλλες επιτροπές, ότι μιλάμε για ένα μοναδικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολλά εξειδικευμένα, ειδικότερα προγράμματα. Θα θέλαμε λοιπόν μια ε, μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση των πόρων. Η γενιά του Εράσμους ε, σημαίνει ότι έχουμε τρία εκατομμύρια νέους που μπορέσαν να υποφοληθούν αυτές τις δυνατότητες στο, ε, στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα μιλάμε για πέντε εκατομμύρια Νομίζω ότι 4 εκατομμύρια είναι ένας λογικός στόχος. Ελπίζω πάντως ότι θα μπορέσουμε να διαθέσουμε το Εράσμο σε περισσότερους νέους της Ευρώπης. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προωθήσουμε γλωσσικές γνώσεις επίσης. Πρέπει να διδάξουμε νέες καριέρες, νέο τρόπο ζωής, άλλες δεξιότητες, μεγαλύτερη αποσχολησιμότητα. Τώρα, μια άλλη προτεραιότητα αφορά ένα συγκεκριμένο τμήμα της συνεχιζόμενης παιδείας, που τον παραγνωρίζουμε καμιά φορά αυτό το τομέα. Αναφέρομαι στις μεταπτυχιακές σπουδές, επίπεδου δοκτορά. Ε, ξέρουμε ότι ο ρόλος των ε, σπουδών στο μεταπτυχιακό επίπεδο μπορεί να ε, προωθήσει την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης. Είναι ζωτικό αυτό για τις κοινωνίες μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε δει εθνή συνεργασία σε αυτό το επίπεδο των σπουδών και διεπιστημονική προσέγγιση. Και αυτό είναι σωστό να περιλαμβάνει όλο τον τομέα της παιδείας από τη στιγμή που φεύγουν τα παιδιά από το σχολείο. Στην Πάντοβα θα έχουμε μία συνάντηση το Νοέμβριο. Στις 21 Νοεμβρίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και θέλουμε να προωθήσουμε την συνεργασία σε αυτόν τον τομέα μέσα στο πλαίσιο των ε, συστάσεων της Υπουργικής Διάσκεψης για τη διαδικασία της Μπολόνια που έγινε στο Βουκουρέστι. Αυτή η διαδικασία της Μπολόνια είναι σημαντική και αξίζει παρακολούθησης. Υπάρχει τώρα ένας ε, βαθμός ε, δημιουργίας προτύπων που σέβεται μεν τη διαφοροποίηση ε, μέσα στο πλαίσιο της Μπολόνιας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τώρα λοιπόν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που πιστεύω ότι θα υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και έχουμε τρία βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η πολιτική μας και τα οποία έχουν διαμορφωθεί μετά από την αξιολόγηση 15 ετών. Καταρχάς πιστεύουμε ότι η τριτοβάθμια παιδεία πρέπει να αναπτυχθεί στην Ευρώπη μία νέα πολιτική αναζωογόνηση στις διαδικασίες της Μπολόνιας βεβαίως και τα καινούργια θέματα, τα νέα θέματα, τα οποία θα ήθελα να παρουσιάσω περιληπτικά. Είναι με αυτά που θα ασχοληθούμε στο μέλλον. Καταρχάς πρέπει το περιβάλλον στο σχολείο να είναι ευχάριστο, ασφαλές και ε, να υπάρχουν τα κατάλληλα κτίρια, η κατάλληλη υποδομή και να προάγεται η υγιεινή ζωή στο πλαίσιο πάντα των σχολείων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να θα οργανώσουμε διάφορες συναντήσεις και ε, σεμινάρια με τις αρμόδιες διευθύνσεις. Το, το δεύτερο, ο δεύτερος προσανατολισμός μας είναι ε, να ενισχύσουμε και να προάγουμε άλλους τομείς ε, μάθησης όπως παραδείγματο χάρη η μουσική, οι γλωσσικές γνώσεις, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, ε, μουσική και γλώσσες λοιπόν, πρέπει η εκμάθηση αυτών να αρχίσει σε νεαρή ηλικία, σε μικρή ηλικία. Ε, πρέπει να αναπτύξουμε τις ε, γλωσσικές δεξιότητες, την, τον, ε, γενικά δηλαδή την ε, παιδεία, ε, τον αλφαβητισμό, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει 24 επίσημες γλώσσες. Και έχουμε και μεγάλες διαφορές μεταξύ μας, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προάγουμε την πολυγλωσσία και να διατηρήσουμε αυτή την διαφορετικότητα. Και τέλος, αυτή την ποικιλομορφία μάλλον. Χρειάζεται να έχουμε πιο στενή, ένα πιο στενό σύνδεσμο, μια πιο στενή διασύνδεση μεταξύ πολιτισμού και παιδείας η Ευρώπη έχει ένα χειροπιαστό αλλά και άειλο, μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά και πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργάζονται αυτοί οι δύο τομείς στενά. Δηλαδή να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ παιδείας και πολιτισμού έτσι ώστε να μπορεί η παιδεία να βοηθήσει τα, τη νέα γενιά να ασχοληθεί σε πολιτιστικούς τομείς, να δουλέψει σε πολιτιστικούς τομείς διότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ αγοράς εργασίας και ε, πολιτισμού. Να ανοίγουν διάφορες δυνατότητες απασχόλησης. Αυτή ήταν μια σύντομη περίληψη των ε, προτεραιοτήτων μας, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, ε, η στενή σχέση μεταξύ αγοράς εργασίας και παιδείας και ε, πολιτισμός και απασχόλησμη πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προάγουμε και να διαμορφώσουμε μία σωστή βάση κατά την Προεδρία μας για την επόμενη εφταετή περίοδο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την κυρία Τζιανίνη για την εισήγησή της και πιστεύω ότι εδώ μας ανοίγεται μια νέα προοπτική, έχουμε μια νέα οπτική γωνιά και νέα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Ιταλική Προεδρία. Πολλές ιδέες, πιστεύω, πολλές από αυτές τις ιδέες τις συμμεριζόμαστε εμείς στο Κοινοβούλιο και θα βοηθήσουμε στην προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων και προσβλέπω σε μια πολύ επιτυχημένη και στενή συνεργασία ε, και μέσα στο Συμβούλιο και μας ε, ε, αρέσει πάρα πολύ η ιδέα και την υποστηρίζουμε τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των Υπουργών Απασχόλησης και των Υπουργών Πολιτισμού έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερή γέφυρα μεταξύ των δύο τομέων μια γέφυρα συνεργασίας. Αυτό μπορεί να στείλει και ένα μήνυμα προς το Κοινοβούλιο, διότι πολλές φορές έχει υπάρξει ένα έλλειμμα κοινή στρατηγικής στο παρελθόν. Θα ήθελα τώρα να δώσω την ευκαιρία να μιλήσουν οι συνάδελφοι μας, τα μέλη μας και θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Κομοντίνη από το ΕΛΚ και κυρία Γκριμπάσκα από τους Σοσιαλιστές. κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας. Έχω μία-δύο ερωτήσεις, θα μιλήσω αγγλικά. Άκουσα τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας και εκτιμώ ιδιαίτερα τα σημεία τα οποία αναφέρεται που αφορούν την ε, μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την απόκτηση διδακτορικού και την πρόθεση προγραμμάτων που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Ε, καταρχάς, ε, τη, τα παιδιά, τους μαθητές οι οποίοι εγκαταλείπουν τη σχολική εκπαίδευση ε, νωρίς. υπουργοί στο παρελθόν μας είχαν υποσχεθεί ότι αυτό το ποσοστό θα μειωθεί σημαντικά και το θέμα αυτό του ποσοστού εγκατάλειψης σχολικής εκπαίδευσης έχει άμεση σχέση με την απασχόληση και με την απασχόληση των νέων, της ανεργίας των νέων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας ε, απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις. Τι προτεραιότητα θα δώσει η τελική προεδρία σε αυτό το θέμα, τι πόρους ε, θα, χρησιμοποιήσει ή θα διαθέσει και τρίτον, εάν η Προεδρία έχει υπόψη συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχύσει ε, την, ε, τρέχουσα, τις τρέχουσες δραστηριότητες που ήδη εφαρμόζονται. Το, όσον αφορά τώρα ε, την, τα, προγράμματα προτεραιότητας για τους νέους, αναφέρατε ότι το έχετε ενσωματώσει στις προτεραιότητές σας και ότι ειδικά στη Μάλτα που είναι η χώρα μου προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ ε, της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων και των ε, νέων και πιστεύω ότι αυτή η στενή σχέση πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω δηλαδή παιδεία και ε, επιχειρηματικός κόσμος επιχειρηματικότητα. Όμως εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, μερικά εμπόδια. Παραδείγματο χάρη, έλλειψη χρηματοδότησης. Ε, μετά, ε, την απαραίτητη εγγυητική διαδικασία για να μπορέσει κανείς να προωθήσει αυτή την συνεργασία. Πώς θα χειριστείτε αυτό το θέμα, θα προωθήσετε αυξήσετε την επιχειρηματικότητα των νέων βεβαίως, αλλά πώς θα συνδέσετε ε, αυτή την προτεραιότητα με την ε, κατάργηση των εμποδίων που υπάρχουν συγκεκριμένα και που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας όταν θέλουν να μπουν στον επιχειρηματικό κόσμο. Ευχαριστώ η Πρόεδρος, ευχαριστώ την κυρία Κομοντίν, κυρία Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων στο θέμα της παιδείας και της ανάπτυξης. Η φιλοσοφία σας ε, την υποστηρίζω θερμά. Μου επιτρέπετε να θέσω ορισμένες ερωτήσεις με τη σειρά που παρουσιάσετε και εσείς τα θέματά σας. Πρώτον, έρευνα. Θα κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας θα ξεκινήσετε μία νέες κατευθύνσεις στην έρευνα, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάμεινο. Την, για την ενίσχυση των πόρων, των χρηματοδοτικών πόρων για την έρευνα, έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Εάν θέλουμε να ε, οικοδομήσουμε μία παιδεία που βασίζεται στην έρευνα, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων και να μην εμπέσουν στις περικοπές του προϋπολογισμού. Δεύτερον, η, η αύξηση της απασχόλησης. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα γιατί θα συζητήσουμε το θέμα της διτής εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους όχι μόνο θεωρητικά να μάθουν αλλά και πρακτικά να ασχοληθούν με ε, μία μαθητεία. Λοιπόν, θεωρητική εκπαίδευση αλλά και πρακτική μάθηση και το τονίζω σε κάθε στάδιο, σε κάθε βασμίδα της εκπαίδευσης, ακόμα και στα μεταπτυχιακά και στις διδακτορικές διατριβές, πρέπει να έχουμε παράλληλα την μάθηση, την πρακτική. Έχουμε μία εξαιρετικά εκπαιδευμένη και ειδικευμένη ε, νεότητα, ε, η οποία δεν μπορεί πρακτικά να απασχοληθεί. Και θα πρέπει αυτός, αυτή, αυτός ο διτός ε, χαρακτήρας της μάθησης και της πρακτικής εφαρμογής για να έχει επιτυχία χρειαζόμαστε μια σταθερή ε, ευρωπαϊκή βάση εκπαίδευση, παιδεία, μάθηση αλλά και πρακτική πρακτική ε, μάθησης έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μία όθηση σε αυτό το διπλό, διτό σύστημα παιδείας. Και θα τονίσουμε και την πολυπολιτισμική διάσταση της Ευρώπης. Μία άλλη, ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ιταλικής Προεδρίας είναι ότι προωθεί μια στενότερη συνεργασία πολιτισμού και ε, οικονομικού τομέα, ε, επιχειρηματικού κόσμου. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να δίνουμε και τις κατάλληλες υποτροφίες, ιδίω για τεχνική εκπαίδευση, ας πούμε οι φοιτητέ των πολυτεχνείων, τα πολυτεχνία, οι τεχνικές σχολές, εκτός από τις κλασικές σπουδέ και τις ανθρωπιστικές σπουδέ, πρέπει να δίνουμε υποτροφίες και για στα τεχνικά ιδρύματα, στα πολυτεχνία. Αν κάποιος ε, φοιτητής ε, ε, που είναι φοιτητής αρχιτεκτονικής μπορεί, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει και φιλοσοφία, να μην αποκλείει το ένα το άλλο. Και επανέρχομαι τώρα και στην, στην επιχειρηματική και οικονομική διάσταση. Εγώ ήμουν υπουργό πολιτισμού στην Πολωνία και ε, είχα ήδη σκεφτεί ορισμένες από αυτές τις ιδέες και ένας μαθητής ε, μετά από το μάθημα μου είπε «Μα τι θέλει αυτή η κυρία, πώς μπορεί αυτή η κυρία να μας βάλει στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ε, εάν ήταν επιχειρηματικό το πνεύμα της ε, δεν θα, θα ερχόταν εδώ να μας ε, διδάξει. Άρα λοιπόν χρειάζεται και εκπαίδευση των δασκάλων, όχι μόνο των μαθητών και των δασκάλων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Η κυρία Κάμερ Μάιερτ. Ευχαριστώ, κυρία πρόεδρε έχετε παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και δεδομένου ότι η Προεδρία διαρκεί μόνο ένα εξάμεινο, ε, είμαστε συνέχεια υπό χρονική πίεση και ιδιαίτερα εδώ στο Κοινοβούλιο το θέμα της παιδείας αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον. Μπορούμε βεβαίως να εκδώσουμε όσες συστάσεις ε, θέλουμε και να δηλώσουμε την προθυμία μας, τη δέσμευσή μας, τις υποσχέσεις μας και ούτω καθεξής. Και όπως είπε και η συνάδελφός μου για τη διτή ε, εκπαίδευση, συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε την ε, εγγύηση των νέων. Εγγύηση για τους νέους. Είναι μία ιδέα προς την οποία έχουμε δεσμευτεί. Δεν διαθέσαμε αρκετά κονδύλια, αρκετές πιστώσεις και τώρα αντιμετωπίζουμε μια τεράστια ανεργία των νέων, ιδίως στα νότια κράτη της Ευρώπης. Χρειάζονται λοιπόν και βελτιώσεις στις υποδομές, τις κρατικές υποδομές, και όλοι πάντοτε τονίζουν το γερμανικό σύστημα εκπαίδευση και μαθητεία και όλοι λένε ότι αυτό πρέπει να το υιοθετήσουμε, είναι πρότυπο κλπ. Αλλά το θέμα το γερμανικό, στη γερμανική παράδοση αυτή της διτής εκπαίδευσης, την οποία εφαρμόζουμε εμείς και δεκαετίας, συμπεριλαμβάνει και την τεχνική τεχνική εκπαίδευση επιτόπου. Δηλαδή, μαθητεία μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στις ε, επιχειρήσεις και το κράτος έχει βεβαίως την ευθύνη της ε, θεωρητικής εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν ε, πληρώνει, δεν χρηματοδοτεί μόνο το κράτος την παιδεία, αλλά χρηματοδοτούν και οι επιχειρήσεις, ο οικονομικός τομέας δηλαδή, αναλαμβάνει τη χρηματοδοτική ευθύνη για την μαθητεία την τεχνική επιτόπου εκπαίδευση. Ε, πολλές φορές Πολλές φορές βεβαίως οι επιχειρήσεις λένε ότι η ιδέα αυτή είναι καταπληκτική αλλά το κόστος θα πρέπει να, να το φέρει όλο το κράτος ή το δημόσιο, η κυβέρνηση δηλαδή. Πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες αλλά το κράτος να πληρώσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε πρακτικά ε, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη απασχόλησης. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μην υιοθετήσουν κυριολεκτικά το σύστημα αυτό ως έχει, αλλά να εξετάσουν καταρχάς πού υπάρχει ανάγκη, πού υπάρχουν τα κονδύλια, ποιες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες και σιγά-σιγά να το εισαγάγουν. Στην προηγούμενη θητεία ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα και με τα, μέσα, με τα οπτικοακουστικά μέσα και την ενημέρωση και τη χρησιμοποίηση των νέων μέσων όταν οι νέοι μας είναι, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, έχουν αυτοπεποίθηση, μπορούν να χειριστούν τα νέα τεχνολογικά μέσα, τα νέα κοινωνικά μέσα, τα οπτικοακουστικά, όλα αυτά ε, και αυτά χρειάζονται μία... Όταν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν όλη αυτή τη τεχνολογία έχουν πολλές δυνατότητες ιδίως στην ε, διαδικασία της Μπολόνιας. Στη Γερμανία και σε όλα κράτη-μέλη πιστεύω ότι εφαρμογή, υλοποίηση ε, όλων αυτών για τα οποία έχουμε παλέψει είναι ελιπέστατη. Πάρα πολλοί φοιτητέ μας ε, λένε ότι έχουν μία υποτροφία Εράσμους την χρησιμοποιούν την υποτροφία αυτή, αλλά γυρίζοντας στην πατρίδα τους δεν αναγνωρίζονται. Οι βασμοί τους δεν, δεν ε, ωφελούνται από αυτήν την διαδικασία του Εράσμους. Τώρα, έχουμε αυτό το αιώνιο πρόβλημα της αμοιβέ αναγνώρισης. Εάν ένα ε, εκπαιδευτικό είδημα δεν αναγνωρίζει ε, τα πτυχία ή τα πιστοποιητικά του άλλου, πώς θα βοηθήσουμε έτσι πρέπει με, με όλες μας τις ε, δυνάμεις και πάλι να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη που υπάρχουν, ε, ε, παρουσιάζουν αυτά τα εμπόδια και αυτά τα προσκόμματα, ότι εμείς δεν δημοσιεύουμε μόνο ιδέες, αλλά είμαστε υπεύθυνοι και για την υλοποίηση οι φοιτητέ μας εάν έχουν την δυνατότητα και την γνωρίζουν ε, ότι αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, αναγνωρίζονται ε, αυτές οι ανταλλαγές οι εκπαιδευτικές θα έχουν και περισσότερο ενθουσιασμό να τις χρησιμοποιήσουν. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ Πέτρα. Ο, η κυρία Τούμ. Ε,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 είναι ένα θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προϋπόθεση παροχής της βέλτιστης παιδείας είναι να είναι πολύ καλό το σχολικό μας σύστημα. Δηλαδή να μην έχουμε μόνο στο νου μας την διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, αλλά και την προστασία των μειονοτήτων, την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης ε, στις μειονότητες, τους Ρωμά ε, ε, και το μόνο ο μόνος δρόμος που, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλου είναι μέσω του Εράσμους. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να προωθήσουμε αυτή την πολυπολιτισμικότητα στο σχολικό σύστημα, όχι μόνο αργότερα. Δεν είναι μόνο η εκμάθηση ξένων γλωσσών, αλλά και η ενσωμάτωση στην παιδεία, ιδίως στη σχολική, όλων των μειονοτήτων. Ο κ. Μαλτέζε. Ευχαριστώ πολύ την Υπουργό για την παρουσία της εδώ και για την παρουσίασή της. Ιδιαίτερα όμως για τον τρόπο τον οποίο ε, υπεραμείνθηκε του προγράμματος ε, Εράσμους. Όπως το έκανε άλλωστε και ο Ιταλός Πρωθυπουργός στο Στρασβούργο όταν παρουσίασε την επερχόμενη Ιταλική Προεδρία. Απ' την άλλη ε, μεριά υπάρχει και η καθημερινή πρακτική, η καθημερινή μάχη την οποία πρέπει να δώσουμε για να προασπίσουμε το Εράσμους. Συνεπώς ε, θα ήθελα να σας ξανακάνω έκκληση κύριε Υπουργέ η Ιταλία να δώσει αυτή τη μάχη συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και να υποστηρίξει τις ε, πρωτοβουλίες της ε, δικής μας ε, Προέδρου η οποία αποφάσισε ότι θα στείλει επιστολή στον κύριο Γιούνκερ για να τονιστεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αρμόδιου για θέματα πολιτισμού επιτρόπου. Ε, Ιταλία αντιπροσωπεύεται με την κυρία Μογκερίνη στην ε, Κομισιόν, αλλά θα ήθελα και η Ιταλική Προεδρία να κάνει το δικό της καθήκον. Βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα οποία είναι λίγο ε, ε, που εκκρεμούν και δημιουργούν αμφιβολίες για παράδειγμα τη δυνατότητα των τραπεζών να δίνει δάνεια σε φοιτητές χρειάζεται μια... Ε, καλύτερο θα ήταν να τους ε, ε χορηγούμε υποτροφίες ε, και όχι δάνεια. Έτσι, γιατί με ένα δάνειο ο φοιτητής μετά τελειώνει τις σπουδές του και χρωστάει. Καλύτερα να του δίνονται υποτροφίες όπως το Εράσμους, μέσω του Εράσμους. και ένα τελευταίο σχόλιο, χωρίς να θέλω να είμαι έτσι επιθετικός ή αριστικός. Ε, η... Μερικές φορές βλέπω ότι υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτά που εξαγγέλει η κυβέρνηση, η Ιταλική κυβέρνηση για το εξάμεινο και την πρακτική στην Ιταλία. Δηλαδή τι γίνεται στην Ιταλία. Υπάρχει ένα έλλειμμα επενδύσεων ε, στον τομέα του πολιτισμού και τη παιδείας τα τελευταία χρόνια. Και βρισκόμαστε αρκετά κάτω του ευρωπαϊκού μεσουόρου. Γενικότερα έχει παρατηρηθεί μια πολιτιστική και οικονομική υποχώρηση στη χώρα μας. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα τα καταφέρει και θα αντιστρέψει αυτή την τάση. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ε, ε παρατηρήσεις Υπουργού ε, διαβάσαμε ότι ε, πέρασατε πολύ ωραίες διακοπές. Ελπίζουμε, χαίρομαστε που σας βλέπουμε εδώ ξεκούραστη κυρία Υπουργέ. Ε, για όσο χρόνο μένει από το Ιταλικό εξάμεινο. Θα πρέπει ασφαλώς να είμαστε επικοδομητικοί. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν βρίσκω καμία ερώτηση που να είναι πραγματικά επικοδομητική. Ε, εγώ έχω σπουδάσει αρχαιολόγος, ε, είμαι, ήμουν ε, δασκάλα, προέρχομαι από την Νότια Ευρώπη όπου οι γυναίκες στην περιοχή μου τουλάχιστον πλήττονται από ποσοστά ανεργίας γύρω στο 45%. Έχω στο μυαλό μου πολύ τους νέους ανθρώπους ιδιαίτερα και κάθε φορά που βλέπω τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παιδεία, το μόνο που παρατηρώ είναι τα απίστευτα αρνητικά νούμερα για την Ιταλία. Τελευταία, κάτω-κάτω στον κατάλογο, σε ό,τι αφορά τους ε, μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχουμε 39.000 λιγότερα άτομα που πήραν πτυχίο από το Πανεπιστήμιο φέτος από σχέση με πέρσι. Ε, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εγκατάλειψης ε, ε, ε, το, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 29% με μέσο όρο 11% ε, μόνο το 55% των φοιτητών πήραν πτυχίο πέρσι τα νούμερα πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστα έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά παχύσαρκων παιδιών, 35% συνολικού αριθμού των παιδιών μας είναι παχύσαρκα. Τι να σας πω κύριε Υπουργέ, ε, η Ευρώπη ε, ασφαλώς πρέπει να είναι μεγάλη ευκαιρία για μας γιατί είμαστε κάτω-κάτω στον κατάλογο, στον πάτο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα κάνει καλά τη δουλειά της η Προεδρία. Οπότε το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πώς αισθάνεστε τώρα να είστε εδώ μπροστά μα και να αντιπροσωπεύετε μια χώρα που είναι στον πάτο τη Ευρώπη. Ε, ποιες είναι οι βέλτιστες ε, πρακτικές που θα ε, μπορέσουμε εμείς ε, το δικό μας σήμα να δώσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόεδρος. Θα δώσω θα δώσω το λόγο στον κύριο Γραμματικάκη, αλλά παρακαλώ πολύ να μην γίνει μια Ιταλο-Ιταλική συζήτηση εδώ πέρα. Ο κύριος Γραμματικάκης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βλέπω εδώ την Υπουργό Παιδείας της Ιταλίας και πολύ σωστά η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό και ιδιαίτερα στο Erasmus Εγώ θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση, κυρία Υπουργέ, ε, και μία ερώτηση. Η γενική παρατήρηση είναι ότι από την πρώτη στιγμή είμαι νέος Ευρωβουλευτής. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο ακούω από όλους τους υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και από τον κύριο Γιούγκερ τη σημασία του πολιτισμού, της παιδείας και όλων των συναφών αρμοδιοτήτων. Όπως όμως λίγο υπονοήσατε κι εσείς με ευγένεια η στο στρασβουργο ακουω απο ολους τους υπευθυνους της ευρωπαικης ενωσης ακομα και απο τον κυριο γιουγκερ τη σημασια του πολιτισμου της παιδειας και ολων των συναφων αρμοδιοτητων οπως ομως λιγο υπονοησατε κι εσεις με ευγενεια τα λόγια από την πράξη έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Υποτίθεται ότι ο πολιτισμός και η παιδεία είναι τα θεμέλια της Ευρώπης, αυτό όμως ε, δεν γίνεται καθημερινή πράξη και ειδικά με τη σημερινή κρίση που ζουν κυρίως οι νότιες χώρες, ε, κάνει τα μεγάλα αυτά λόγια να φαίνονται με μια αρχαία ρίση έπεα και θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι στη διάρκεια της Προεδρίας σας, γιατί δείξατε ένα συγκροτημένο σχέδιο για την παιδεία, να εξαντλήσετε όλο το δυναμισμό σας για να αποκτήσει η παιδεία τουλάχιστον κάποια εγκύτερη απόσταση προς τα μεγάλα λόγια. Η ερώτησή μου τώρα, σε όλο σας το συγκροτημένο αυτό σχέδιο, αλλά και πριν από αυτό στις διαδικασίες που έχω ακολουθήσει, Υπάρχει ένα παλιό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έλεγα διαρκώς οξύνεται με την οικονομική κρίση αλλά και με τη νέα φορά της εποχής. Αυτή είναι κυρία Υπουργέ ο αργός αλλά σαφής παραμερισμός των λεγόμενων ανθρωπιστικών σπουδών σε όλα τα σχέδια ή τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η φιλοσοφία, η ιστορία, οι κοινωνικές επιστήμες ακόμα και η θεωρητική φυσική έχουν μία τάση υποβαθμίσεως στο όνομα της επιχειρηματικότητας ή των αγκαίων ε, ε, απασχόλησης και διάφορα πράγματα που πολλές φορές δεν είναι αλήθεια. Να σας τονίσω ότι είμαι καθηγητής της φυσικής, άρα θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένος γιατί οι θετικές επιστήμες είχαν μεγάλη, αν θέλετε, τόνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν χαθούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, αυτό είναι το ερώτημά μου, ένα σχόλιο απλό περιμένω, τότε ένας από τους θεμέλιους λίθους ε, της Ευρώπης θα έχει οριστικά απολυστεί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Γραμματικάκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ που υπογραμμίσατε ρόλο της Ιταλικής ε, Προεδρίας ε, στην ε, εδραίωση της σύνδεσης ανάμεσα στον πολιτισμό και την παιδεία. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά καμπανάκια σήμερα και πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά θα ταξίδευα στην Ιταλία πρώτα απ' όλα για πολιτισμό και για άλλους λόγους, αλλά κυρίως για κουλτούρα και πολιτισμό. Μία σύσταση, αν θέλετε αλλιώς μία μου επιφύλαξη. Αναφερθήκατε στην ανάγκη αναθεώρησης των στόχων της ε, στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020. Προσωπικά δεν θα σύστηνα αυτό να γίνει με έναν τρόπο δημόσιο. Γιατί, γιατί η στρατηγική στόχη της Ατζέντα 2020 είναι πολύ καλή. Για την τριτοβαθμία εκπαίδευση, ας πούμε, το 50% των πολιτών να φτάνουν στην τριτοβαθμία εκπαίδευση είναι ένας στόχος της Ατζέντα 2020. Ο άλλος στόχος ε, είναι ε, πρόορη εγκατάλειψη ε, της σχολικής ε, κατάρτισης ε, σε ποσοστό μικρότερο του 10%. Νομίζω ότι ελπίζω ότι δεν θα αναθεωρήσετε αυτούς τους στόχους ούτε και θα το σύστηνα γιατί το Εράσμους έχει ευθυγραμμιστεί με αυτούς τους στόχους και με κάποιους άλλους ε, πιο δευτερεύοντες, ε, πιο επιμέρους. Εγώ θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω μία ιδιαίτερη δραστηριότητα που είναι πολύ σημαντική, την στήριξη της ε, γλωσσομάθειας, της γλωσσικής εκπαίδευσης. Σε, συνδυασμό με ε, επισκέψεις. Θα πρέπει και οι δάσκαλοι γλωσσών, και οι δάσκαλοι, και οι καθηγητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές να εκπαιδευτούν στις γλώσσες. Η Ιταλία δεν είναι τελείως στον πάτο. Το 2013 είδαμε τα αποτέλεσματα του Πίζα και είδαμε ότι η Ιταλία είναι καλύτερη από την Τσεχική Δημοκρατία. Ε, για παράδειγμα σε θέματα ε, ε, του αγάπης προς το σχολείο. Για παράδειγμα λέω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε εμείς στη χώρα μας βέβαια. Θα ήθελα και τα δικά μας παιδιά να αγαπάνε το σχολείο τους περισσότερο. Αυτό είναι ένα όμως εσωτερικό μας ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ για την ε, πρωτοβουλία να αναθεωρήσετε την διαδικασία της Μπολόνια. Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα, απαραίτητο όμως. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να γίνουν τα καλύτερα στον κόσμο. Και πρώτα βέβαια πρέπει να εντοπίσουμε τα εμπόδια. Καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες σας λοιπόν, εκ βάθους καρδίας και τέλος θα σας πρότεινα να μην αλλάξετε τους βασικούς μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δίνουν μια ασφάλεια. Το επαναλαμβάνω αυτό το είπα και προηγουμένω. Δίνουν ασφάλεια και προβλεψιμότητα στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε. Ο χρόνο ε, πιέζει λίγο. Έχουμε ήδη πάρει μια καθυστέρηση και έχουμε πέντε ακόμα μιλητέ στον κατάλογο. Και κλείνω τον κατάλογο αυτή τη στιγμή με αυτά τα πέντε ονόματα. Παρακαλώ πολύ να είστε σύντομοι και σύντομες, έτσι ώστε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Κύριε Βόρτ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ θετική ήταν η παρουσίασή σας και σαφής και συνεκτική. Αυτά τα στοιχεία της συνοχής ε, μας έλειπαν και είναι και ένα πρόβλημα που μας δυσκολεύει ιδιαίτερα στο να προάγουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά που άκουσα σχετικά με την ε, κατάργηση των εμποδίων ε, που, που αντιμετωπίζουν οι νέοι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι νέοι και το μέλλον τους και πραγματικά πρέπει να, να μπορούν να ξεπεράσουν πολλά από τα υπάρχοντα εμπόδια. Αναφέρομαι τώρα, ε, επειδή εκεί έχω εργαστεί, στους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες ε, είναι και επιχειρηματίες, ασχολούνται με επιχειρηματικά θέματα. Ο Πίτερ Μπρουκ, ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ε, έχει πολλές φορές μιλήσει για αυτό το θέμα και πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να δημιουργήσουν θαυμάσια πράγματα μέσα σε έναν άδειο χώρο. Μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε την επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, με την καλλιτεχνική ε, έκφραση. Είναι μια θαυμάσια ιδέα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ε, χρειάζονται χώρο να, παίξουν και δεν εννοώ παιχνίδια, ενώ να πειραματιστούν, να διαμορφώσουν, να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της επιχειρηματικότητας θέλω να περιλάβετε και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, διότι ε, το επιχειρηματικό πνεύμα μπορεί πολλές φορές να είναι πολύ εγωιστικό και ε, πολλές, σε πολλές περιπτώσεις μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Επιχειρηματίες και επιχειρηματικό πνεύμα έχουν και τραπεζίτες, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει και την κοινωνική πτυχή είναι πολύ πιο σημαντικό, πολύ πιο ενθαρρυντικό όταν ε, το επιχειρηματικό πνεύμα έχει και μια κοινωνική διάσταση. Όσον αφορά τώρα την, ε, τα ψηφιακά μέσα, την ψηφιακή μας εποχή, έχουμε καθήκον να προάγουμε τη χρήση των δυνατοτήτων αυτών και στον λιγότερο ανεπτυγμένο κόσμο ε, ο Σουγκάτρα Μήτρα ήταν δάσκαλός μου, ο οποίος είναι καθηγητής και ειδικό στην τεχνολογία των computers στην Ινδία και έχει κάνει προβολές μέσω κομπιούτερ στο, σε τείχους, σε, σε νέους ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ έρθει σε επαφή με την τεχνολογία αυτή ούτε την είχαν ποτέ χειριστεί. Μην είμαστε λοιπόν υπερόπτες και μιλάμε συνέχεια για ψηφιακή τεχνολογία, τον ξέρουμε ότι σε άλλα μέρη του κόσμου ούτε καν υπάρχει, είναι γνωστή. Εν συνεχεία, η δυνατότητα συμμετοχής ε, των κοινοτήτων, της κοινότητας. Ε, έχω ασχοληθεί σε διεθνή κλίμακα ε, μέσω ενός κέντρου για την συμμετοχή νέων και κοινοτήτων σε, προγράμματα τα οποία είναι διεθνή. Δηλαδή να ξεπεράσουμε την τοπική μας κοινωνία και να επεκταθούμε και διεθνώς. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ ο κύριος Διάκονο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε από την κυρία Υπουργό είναι πάρα πολύ καλά νέα, διότι μας μίλησε για συγκεκριμένα θέματα τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς. Όπως και η κυρία Λιμπάτσκα, εγώ και εγώ ε, μία, ένα δικό μου έτοιμα. Η χώρα μου, η Ρουμανία, στη Ρουμανία προσπάθησα να χτίσω ένα σπίτι και προσέλαβα τους τεχνίτες, ε, τους οικοδόμους, ε, τους μπογιατζίδες, όλοι αυτοί που χρειάζονται. Κάποια στιγμή ήρθε ένας νέος λοιπόν και σε μένα και είπε «Κύριε Μίρτσα, σε παρακαλώ βοήθησέ με να βρω μία δουλειά. Γιατί δεν θέλω να εργαστώ πια. Αυτό δεν βγαίνει σωστά όταν μεταφράζουμε τα ρουμάνικα, αλλά στα ρουμάνικα, φαίνεται στη ρουμανική γλώσσα, υπάρχει μία διαφορά μεταξύ εργασίας και δουλειάς. Αυτό που ζητούσε ο άνθρωπος είναι, είναι μία εργασία καλύτερη από τα οικοδομικά. Αυτό που ήθελε λοιπόν δεν είναι περισσότερο λεφτά, γιατί λεφτά έβγαζε στην οικοδομή, αλλά ήθελε κύρος, κύρος. Και η δουλειά αυτή της οικοδομής δεν έφερνε το κύρος που ήθελε ο άνθρωπος και ήθελε μια εργασία καλύτερη. Όταν λοιπόν μιλάτε για επιχειρηματικότητα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις νοοτροπίες. Η νοοτροπία που υπάρχει είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. πώς βλέπει κανείς τη, δουλειά, την εργασία. πολλές φορές η σχέση μεταξύ σχολείου και οικογένειας, σχολείου και κοινωνίας είναι πολύ σημαντική ε, διότι εκεί διαμορφώνονται απόψεις που πολλές φορές είναι πρόβλημα στην εποχή μας. Γιατί το τονίζω. Αυτή η σχέση σπιτιού, ε, παιδείας, ε, κοινωνίας, οικογένειας εάν δεν λειτουργεί σωστά, στη Γερμανία, πούμε, τα προβλήματα είναι σε μεγάλο ποσοστό ξεπερασμένα. Ε, συνεχώς αναζητούν οι νέοι ένα επάγγελμα μέσω δηλαδή της παιδείας το οποίο είναι ε, ε, τιμητικό, έχει δηλαδή κύρος, έχει μία, ε, μία έγλη, μία έγλη. και γι' αυτό θα πρέπει να εξαφανίσουμε αυτήν την νοοτροπία, να, καταργήσουμε αυτή την νοοτροπία διότι είτε κάποιος κάνει διδακτορικό, είτε ένας νέος εγκαταλείπει το σχολείο και ακολουθεί ας πούμε μια εγκληματική πορεία και τα δύο προβλήματα μας απασχολούν. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ένα από το άλλο. Ο κύριος Μοργάνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ. Να τονίσω και εγώ μερικά σημεία μετά από την έξοχη εισήγησή σας. Πρέπει να κάνουμε συνεχώς μία αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, διότι όπως είπατε, αποκτάτε γνώση, αλλά χρειάζεται συνεχώς να, να ανανεώνουμε, να επικαιροποιούμε τη γνώση αυτή. Αναφέρεστε σε μια σειρά πρωτοβουλειών που δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν ε, άμεσα και αυτό ισχύει βεβαίως και για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Εκεί πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, τα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα και η παιδεία και η έρευνα σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ανεργίας των νέων. Η στην αντιπροσωπεία που είμαι θα ε, δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών διότι κάθε κράτος κάνει τα δικά του ενώ εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία και τη λεγόμενη συνέργεια στα προγράμματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάποιος που, που είναι στο σχολικό σύστημα και καθ' όλη τη διάρκεια της παιδείας του θα πρέπει να καταλάβει ότι η παιδεία δεν εξασφαλίζει διαβίου απασχόληση, δηλαδή μία δουλειά την οποία θα πάρει δεν θα τον εξασφαλίσει διαβίου, διότι αυτό τώρα είναι μία πραγματικότητα της ζωής. Και εάν δεν καταλάβουν ότι δεν είναι εξασφαλισμένοι για όλη τους τη ζωή στην πρώτη εργασία που θα πάρουν, ε, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα μελλοντικά εμπόδια. Σας ευχαριστώ επίσης που τονίσατε την τεχνική και πρακτική μάθηση. Βεβαίως εμείς δεν έχουμε φτάσει το επίπεδο της Γερμανίας, αλλά πιστεύω ότι η κατάσταση βελτιώνεται σε μας και θα υπάρχει οπωσδήποτε ένα οικονομικό όφελος εφόσον ε, ε, αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η πρακτική μάθηση, η πρακτική παιδεία. Επίσης ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε μια πιο στενή σχέση μεταξύ οικογένειας, παιδείας και εργασίας, ε, της, ε, της απασχόλησης. Πιστεύω ότι τα επίπεδα της τριτοβάσμιας, το επίπεδο της τριτοβάσμιας εκπαίδευσης και τα διδακτορικά θα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον, διότι μας δίνεται η δυνατότητα να ανταγωνιστούμε διεθνώς και να προβάλλουμε την Ευρώπη ε, ως, σύγχρονη ε, και να, να ξεπεράσουμε τις, ε, τις αγγυλώσεις του παρελθόντος. E και βεβαίως να προωθήσουμε και την εφαρμοσμένη έρευνα αλλά και τις ανθρωπιστικές κλασικές σπουδές διότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με, τα κατάλληλα, με τις κατάλληλες πιστώσεις. Αν δεν έχουμε τα, κατάλληλα, ε, τα αναγκαία χρήματα, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πάρα πολλοί διαμαρτύρονται για τις περικοπές στο πρόγραμμα Εράσμους. Οπωσδήποτε πρέπει να αντιδράσουμε στις περικοπές αυτές, διότι έχω, ε, ε, υπάρχει συμφωνία στο να αντισταθούμε σε αυτές τις περικοπές. Βεβαίως πρέπει να τηρήσουμε τον προϋπολογισμό μας μέσα στο σύμφωνο σταθερότητος, αλλά παρόλα αυτά. Ο κύριος Γλέζος. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ζητάω συγγνώμη διότι λόγια ανυπέρβλητη από τη θέλησή μου με ανάγκασαν να μην είμαι από την αρχή στη συνεδρίασή σας. Μπροστά στην ε, μαύρη μαυρίλα που έχει πλακώσει την ε, Ευρώπη, μαύρη σαν καλιακούδα όπως λέει ένα δύστιχο ελληνικό, έχω να σας ανακοινώσω ένα πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Είναι οι έρευνες που γίνονται και που παρουσιάζουν τον τύμβο της Αμφίπολης στην Ελλάδα. Δυστυχώς η επισήμανση του πολιτισμικού αυτού στοιχείου έγινε από το 2009. Πέρασαν πέντε χρόνια για να πιστεί η ελληνική κυβέρνηση να δώσει τα χρήματα να αρχίσουν οι ανασκαφές το πολιτισμικό αυτό στοιχείο δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Πρόκειται για δημιούργημα του δεύτερου πολιτισμού της Ευρώπης. Πρώτο υπήρξε ο κυκλαδικός πολιτισμός και ακολούθησε ο μικυναϊκός και είναι δείγμα του μικυναϊκού πολιτισμού. Απαιτούνται όμως αρκετά χρήματα για την ανασκαφή αρκετά χρήματα για τη στήριξη όλης της εργασίας, ειδικό υπόστεγο, ειδικά χρήματα για τη διατήρηση του χώρου, όσοι γνωρίζουν από αυτά τα θέματα πρέπει να πούν και στους άλλους ότι όταν ένα μάρμαρο βγει από τον κρυψώνα του μπορεί αμέσως να ασβεστοποιηθεί και χρειάζεται να διατηρήσουμε το μνημείο όπως έχει. Υπάρχουν τρία κοινοτικά ταμεία τα οποία θα μπορούν να επέμβουν και να δώσουν τα χρήματα για τη συνέχιση ανασκαφής, για την υποστήριξη ανασκαφής, για τη διατήρηση των ευρημάτων και για την αξιοποίηση του πολιτισμικού αυτού μνημείου με το ίδιο πάθος θα μιλούσα και ακόμα περισσότερο εάν υπήρχε ένα παρόμοιο πολιτισμικό στοιχείο πάλι χάρη στην Ιταλία μια νέα πομπιεία με το ίδιο πάθος για οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης. Λυπούμε που ως Έλληνας βρίσκεται αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα και είμαι υποχρεωμένος να το υποστηρίξω. Αλλά εάν θέλουμε μια Ευρώπη του πολιτισμού, εάν θέλουμε μια Ευρώπη όπως υπόθηκε εδώ να μελετηθούν οι γλώσσες και όλα τα σχετικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό το μνημείο του πολιτισμού. Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Grazie onorevole per questo richiamo. Onorevole Ευχαριστώ κύριε Γλέζο. Um, uh, Πρέπει να πω ότι χάρηκα πολύ για την παρουσίαση που έκανε η Ιταλή υπουργό. Uh, πιστεύω ότι έχετε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για τους επόμενους λίγους μήνες που σας μένουν και ελπίζω να τα καταφέρετε γιατί πραγματικά ε, το πρόγραμμα σας αξίζει. Με αυτό το κοκτέιλ λοιπόν απασχόληση, παιδεία και τα λοιπά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις οικονομικές στρατηγικές που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έρχομαι σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα μέτρα λιτότητας. Μόλις βγαίνουμε από το τουνέλι. Έχουν υπάρξει όμως ζημιές κατά τη διαδρομή αυτή στην κρίση. Μεγάλη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και χαίρομαι πολύ κυρία Υπουργέ που μιλήσατε πολύ για αυτό το θέμα. Ένα σημείο δεν τονίσατε, θα έλεγα, ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν οι οικονομικές ε, στρα στρατηγικές ε, και δεν υπάρχει ταυτισή των δεξιοτήτων. Υπάρχουν δηλαδή θέσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν δεξιότητες ε, ε, για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Ο χώρος των, της, των, της επικοινωνίας και της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ένα καλό παράδειγμα. Δεν προσελκύει αρκετούς φοιτητές, ίσως είναι θέμα Μάρκετινγκ είναι ίσως θέμα τρόπου ε, ανατροφής των παιδιών. Ε, είναι σημαντικό όμως να ασχοληθούμε με τον ψηφιακό χώρο γιατί είναι το μέλλον. Η αγορά εργασίας δεν βρίσκει τους σωστούς ε, να απασχολήσει. Η Προεδρία λοιπόν τι θα κάνει για να βελτιώσει αυτό το θέμα αυτόν τον τομέα της παιδείας. Τι μέτρα θα ληφθούν τώρα και για τα ανώτερα παιδεία ε, επίπεδα εκπαίδευσης πάντα μέσα στην ψηφιακή εποχή. Ε, ωραία. Μ' αρέσει η επικέντρωση στην επιχειρηματικότητα. Ήμουν, ε, είμαι, ε, ακόμη ίσως επιχειρηματίας. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Είναι σημαντικές οι σπουδές και θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς προτείνεται για τις σπουδές για την επιχειρηματικότητα, διότι ουσιαστικά δεν μπορείτε να μάθετε την επιχειρηματικότητα όπως μαθαίνετε τη λογιστική. Είναι μία στάση ζωής, είναι μία ανάληψη κινδύνου, ε, δεν γεννιέσαι βέβαια με αυτά, αλλά δέχομαι ε, ότι είναι σε αυτός ο τομέας, αλλά θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι θα το κάνετε. Μίλησα πολύ, το αντιλαμβάνομαι. Ε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θέλω να μάθω λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την προσέγγιση της επιχειρηματικότητας. Ευχαριστώ πολύ που καταλαβαίνετε τους περιορισμούς μας. Ε, η συζήτηση ήταν πραγματικά πολύ ζωντανή. 13 ε, ομιλητές πήραν το λόγο μετά τις ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις της Υπουργού. Θα δώσουμε στην, δώσαμε ήδη στην Υπουργό ένα αντίγραφο της μελέτης για τη διτή εκπαίδευση που περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από σύγκριση των, της πραγματικότητας σε διάφορες χώρες, ε, πολύ σημαντικά για το μέλλον. Ε, ε, θα δώσω τρόπο στην Υπουργό και καλωσορίζω τη Γενική Διευθύντρια Πολιστικής Κληρονομιάς που είναι εδώ μαζί μας. Ε, Υπουργός, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν αφού τις ομαδοποιήσω όσο μπορώ. Καταρχήν κυρία Κομοντίνη μίλησε για την πρόορη εγκατάλειψη ε, της σχολικής εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό πρόβλημα και είχε άμεση σχέση με τα όσα είπα στην αρχή της παρουσίασής μου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προσόντα που παρέχονται από τα σχολεία μας θα είναι ένα όπλο για να, ε, για να καταπολεμήσουμε την πρόορη εγκατάλειψη. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια και στα ανοιχτά σχολεία. Τώρα για την επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να άρουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να μπουν στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Οι εθνικές, ε, είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών, αλλά οι εθνικές ε, πρακτικές ε, ίσως είναι ένας καλός τρόπος να δούμε το θέμα, δηλαδή αυτές οι εθνικές πρακτικές να τις ε, καταστήσουμε κοινό κτήμα. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, να δοθούν κίνητρα στα πανεπιστήμια προκειμένου να εφαρμόσουν πολιτικές κινητικότητας όχι μόνο στο πλαίσιο του Εράσμους αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και εκεί μπορούμε να διδαχθούμε από τις βέλτιστες εθνικές πρακτικές. Κύριε Λιβέτσκα, σας ευχαριστώ πολύ για την σφαιρική σας προσέγγιση. Μιλήσατε για την ε, επιστημονική έρευνα, για την οποία μίλησα και εγώ. Έχει άμεση σχέση με, το, με τα όσα λέμε σήμερα. Εκπαίδευση και επιμόρφωση. Και εκεί συμφωνώ μαζί σας, τα όσα είπατε. Νομίζω ότι όλη η Επιτροπή καλεί την ε, Κομισιό να διασφαλιστεί να δυσφαλιστούν τα κονδύλια στα διάφορα προγράμματα σχετικά με τον ε, πολιτισμό και την παιδεία. Ο πρόεδρος Κομισιόν, ο κ. Γιούνκερ, ε, θα καταρτήσει το στρατηγικό πλάνο για την ε, κατανομή των κονδυλίων. Όμως το σημαντικό είναι σαφές η διτή εκπαίδευση και η η εκπαίδευση ε, με εναλλαγή, εναλλαγή η οποία πραγματικά αποτέλεσε αντικείμενο και άλλων παρατηρήσεων. Η επιχειρηματικότητα και η αυτοεπιχειρηματικότητα επίσης είναι θέματα που πρέπει να υποστηριχτούν πολύ σοβαρά. Και η κυρία Ward το ανέφερε. Θα επανέλθω όμως σε αυτά που είπε η κυρία Ward αργότερα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στην θεματική εκπαίδευση. Θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης. Κύριε Κάμοβερτ. Ε, μίλησε για την ανάπτυξη των ε, πολιτικών σε ε, εκπαίδευσης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η διτή εκπαίδευση είναι εκεί που η εκπαίδευση και η εργασία συνδέονται μεταξύ τους. Η εγγύη στην νεότητα στην νεολαία συγγνώμη, ε, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς. Και νομίζω ότι οι επιχειρήσει πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στην Ιταλία ε, καταρτήσαμε ένα νέο σύμφωνο εκπαίδευσης ε, που εμπλέκει πολλούς φορείς και μέρη της κοινωνίας. Ε, μετά, τα νέα μέσα, οι νέες τεχνολογίες και τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν οι νέοι, να αποκτούν οι νέοι ε, στις νέες τεχνολογίες, τα νέα μέσα, η Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στην Ιταλία και αυτό θα πρέπει να κάνουν και όλα τα κρατημέλη. Αναλαμβάνουμε πολλές πρωτοβουλίες έτσι ώστε μέσα στα σχολεία να δίδεται εκπαίδευση, επιμόρφωση σε νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές και οι φοιτητές και προσπαθούμε επίσης να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Θα πρέπει να τους προετοιμάζουμε για αυτήν την ε, επανάσταση που πρόκειται να έρθει. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε πολύ δραστήριοι όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στα πανεπιστήμια γιατί στα πανεπιστήμια μερικές φορές έχουμε δει επιφυλάξεις. Και ο στην προηγούμενη θητεία είχε κάνει μια χρήσιμη πρόταση για αυτό το θέμα. Η κυρία Τούμ μίλησε για την ε, σημασία των γλωσσών και της ε, πολιτιστικής ε, ποικιλομορφίας, μίλησε για τις μειονοτικές γλώσσες, πολιτισμός και γλώσσα πάνε χέρι-χέρι και υποστηρίζει το ένα το άλλο. δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ε, γλωσσική ποικιλομορφία στα προγράμματά μας. Το Εράσμος είναι εμβληματικό πρόγραμμα, αλλά η ιδέα αυτή των, της πολυγλωσσίας θα πρέπει να εισαχθεί και στα σχολεία. Και έχει ήδη γίνει, τουλάχιστον στην Νότια Ευρώπη, στην Ιταλία, ε, το έχουμε συνειδητοποιήσει και το συνειδητοποιούν και οι νέοι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές προκειμένου να, και συνολικά η ε, κατάρτιση να είναι πολυπολιτισμική ή η εκπαίδευση να είναι πολυπολιτισμική. Ο κύριο Μαλτέζε ε, ζήτησε από την Ιταλική Προεδρία να ε, συμμετάσχει ενεργά και όχι μόνο στα λόγια στην μάχη για την εξασφάλιση επαρκών κονδυλίων για τα προγράμματα κινητικότητας και επίσης να προσπαθήσουμε, μας είπε, να συνδέσουμε τον πολιτισμό με την παιδεία. Ε, η Προεδρία θα υποβάλει τη δική στρατηγική, αλλά πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν το καθήκον του σε εθνικό επίπεδο. Η Ιταλία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εσωτερική πολιτική, αλλά δεν είναι ο χώρος για να τη συζητήσουμε. Ε, ε, πρόσφατα ξεκίνησαν συζητήσει σε εθνικό επίπεδο, επί τη βάση ενό εγγράφου που υπέβαλε η Ιταλική κυβέρνηση. Δεν θα το συζητήσουμε όμω εδώ. Ε, η κυρία Αντινόφη που ε, παρουσίασε κάποια στοιχεία για το που βρίσκεται η Ιταλία στους διεθνείς ε, πίνακες κατάταξης. Ε, όμως να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας αν δείτε πόσοι Ιταλοί έχουν υποβάλει αιτήσει για χρηματοδότηση. Ε, θα σας εκπλήξουν τα στοιχεία. Εθνικά μας ε, θέματα δεν θέλω να τα συζητάμε εδώ. Αλλά έχουμε ήδη ξεκινήσει διαβούλευση με όλη την κοινωνία επί τη βάση ενός εγγράφου που παρουσιάστηκε χτες στη Ρώμη ε, για θέματα εκπαίδευσης. Τώρα, κύριος Γραμματικάκης. Ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε ε, ως επιστήμον που είστε σε, στις ε, θετικές ε, επιστήμες και στις ανθρωπιστικές σπουδές και επιστήμες. Είναι αλήθεια ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι προκλήσεις του, της στρατηγικής 2020 ε, είναι σαφής. Λέει η στρατηγική ότι θα πρέπει και οι δύο αυτές πτυχές και οι θετικές ε, και οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα πρέπει να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο για να λυθούν τα προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική μας κληρονομιά έχει άμεση σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Και ένας από τους στόχους του εξαμήνου μας είναι η προστασία αυτής της πολιτικής κληρονομιάς, όπως το είπα, που σίγουρα πρέπει να περάσει μέσα και από τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή τις ε, θεωρητικές επιστήμες. Ε, μετά, θα, είμαστε, θα διατηρήσουμε τους στόχους του, της στρατηγικής 2020. Ε, είναι φιλόδοξοι, αλλά δεν πρόκειται να τους αλλάξουμε. Ε, η Προεδρία στηρίζει, για παράδειγμα, την ε, γλωσσική εκπαίδευση. Η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια γλώσσα. Ε, η έκθεση Μαλούφ από ό,τι θα θυμάστε και εσείς της προηγούμενες αιτίας του Κοινοβουλίου προέβλεπε δύο γλώσσες συν μία. Και δεν μιλούμε για μια απλή εκμάθηση της γραμματικής του λεξιλεγίου, η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι ένα ολόκληρο πολιτιστικό ταξίδι. Είναι μια περιπέτεια. Κυρία Ward, μίλησε για την ανάγκη να αρθούν κάποια εμπόδια την ε, ε, στηρίζω, την άποψή της ζητάει να δούμε με πιο ευρύ τρόπο το θέμα του επιχειρηματικού πνεύματος να μιλήσουμε για το κοινωνικό επιχειρηματικό πνεύμα, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ε, οι κοινωνικές, ε, μάλλον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο που περιλαμβάνει και τις τέχνες και τον πολιτισμό γενικότερα. Με τη δημιουργία καινούριων απτών ε, μοντέλων ε, επιχειρηματικότητας. Ένας ε, νέος καλλιτέχνης για παράδειγμα ε, να ε, μπορεί μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας να προβάλλει την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Έχω στο μυαλό μου το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ ε, στην Αγγλία. Κύριε Διακόνου, μιλήσατε για την σημαντική, μια σημαντική διάκριση ε, ε, μεταξύ ε, του επαγγέλματος και της εργασίας της εργασίας και της δουλειάς μιλάμε για ένα στόχο απασχόλησης με πραγματική ποιοτικέ θέσει εργασία, με δουλειά, με εργασία αξιοπρεπή που θα δίνει χαρά και θα γεμίζει τους ε, εργαζόμενους. Το είπα και εγώ στην παρέμβασή μου σήμερα το πρωί. Κύριε Μοργκάνο. Ευχαριστούμε πολύ Ε, που μοιράζεστε, συμμερίζεστε μάλλον πολλά από αυτά που είπα και εγώ συμφωνώ με την έκκληση που κάνατε περί της επαρκούς χρηματοδότησης που χρειάζονται οι, ε, τα φιλόδοξα σχέδιά μας Θα συμφωνήσω μαζί σας επίσης το ότι θα πρέπει να δώσουμε όλο και περισσότερη σημασία, να δίνουμε όλο και περισσότερη σημασία στα διδακτορικά, τόσο θεωρητικές όσο και στις θετικές επιστήμες. Τα διδακτορικά δεν δίνουν απλώς γνώση, ανοίγουν πόρτες και παράθυρα ε, και στον κόσμο της εργασίας διότι τα διδακτορικά θα πρέπει να συνδεθούν με τις επιχειρήσεις ε, και μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά τεχνικά, τεχνολογικά και άλλου τύπου ερωτήματα. Κύριε Γλέζο, ο κύριος Γλέζος αναφέρθηκε στη χώρα του στο σημαντικό παράδειγμα της Ελλάδας ε, στις αρχαιολογικές εξκαφές έτσι ώστε να μην χαθεί όχι μόνο η ελληνική ιστορία αλλά και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί πράγματι η Ευρώπη εδράζεται στην αρχαία Ελλάδα πολιτιστικά. Οι Έλληνες δημιούργησαν μια κοινή ταυτότητα για την Ευρώπη μπροστά στους Πέρσες και απέναντι στους Πέρσες. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στι ανθρωπιστικές σπουδέ και ιδιαίτερα ακόμα περισσότερο στην αρχαιολογία. Τέλος, κύριε Μίτση. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Ε, η Υπάρχει πράγματι μια διαφορά στη, στα προσόντα τα οποία έχουν οι φοιτητέ ε, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ένα, ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα προσόντα και στο τι ζητάει η, βιομηχανία, η, η αγορά εργασίας. Θα πρέπει αυτό το χάσμα να το άρουμε. Χρειάζεται προσπάθεια και από εμά αλλά και από τι ίδιε επιχειρήσει. Και οι επιχειρήσει θα πρέπει να υπερβούν αυτό το χάσμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, ε, μια ανάγκη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις να κάνουν μια προσπάθεια να μειώσουν αυτό το χάσμα. με προγράμματα πολύ επιστημονικά, τα οποία δεν θα εστιάζουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μόνο σε μία συγκεκριμένη δίκευση, αλλά θα καλύπτουν ένα ευρύτερο μαθησιακό φάσμα. Η επιχειρηματικότητα, ε, από την άλλη μεριά, είναι ένας τύπος συμπεριφοράς. Ε, η, μια επιχείρηση δεν περιορίζεται σε μια ε, τεχνική. Δεν είναι μια τεχνική και γι' αυτό λόγο και δεν μπορεί να ε, αποτέλεσε αντικείμενο ενό εκπαιδευτικού προγράμματο μόνο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρο. Που ε, απαντήσατε ενδελεχώ σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και Έχουμε προγραμματίσει πολλές άλλες εκδηλώσεις, έχουμε μια πλούσια ημερήσια διάταξη, ένα πλούσιο πρόγραμμα και προσβλέπουμε στενή συνεργασία με πολλούς άλλους συναδέλφους από την Ιταλική Προεδρία. Σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Υπουργέ για τις απόψεις σας και πιστεύω ότι για τον προϋπολογισμό 2015 θα παρουσιάσετε και τις δικές μας απόψεις. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη μας να παραμείνουν στην αίθουσα μετά την αποχώρηση της κυρίας Υπουργού, διότι θα έχουμε την παρουσίαση μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης. Δίνω ένα αντίγραφο της μελέτης αυτής στην κυρία Υπουργό. Ε, είναι η διτή εκπαίδευση και ως Ιταλίδα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αμέσως με την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Ωραία λοιπόν. Θα ε, ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με την παρουσίαση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ε, μελέτης. Η κυρία Ουλίτσνα θα μας την παρουσιάσει και οι συντονιστές αποφάσισαν να στείλουν μία επιστολή στον πρόεδρο Ιούνκερ ε, ζητώντας να εξασφαλίσει ότι ο επόμενος Επίτροπος Πολιτισμού θα έχει ένα ολοκληρωμένο ε, ντοσιέ που θα περιλαμβάνει και δημιουργικές, δημιουργική απασχόληση και συναφή δραστηριότητα που εμπίπτουν στη δική μας ε, σφαίρα ενασχόλησης. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δούμε τη σύνθεση της νέας επιτροπής. Ε, όπως είπε και ο κύριος Μαλτέζε. Η κυρία Ολίτσου να έχει το λόγο. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω σήμερα εδώ τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης την οποία εκφωνήσαμε, την οποία μας ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει τίτλο «Δυτή εκπαίδευση γέφυρα πάνω από θολά νερά» με ερωτηματικό στο τέλος της φράσης. Υπάρχει χρονική πίεση, οπότε θα είμαι σύντομη διότι έχετε και την, την ε, ε, μελέτη αυτή ε, στο φάκελό σας. Ε, μας ζητήσαν λοιπόν να αναλύσουμε διαφορετικά μοντέλα διτής εκπαίδευσης και βασικά την εκπαίδευση στην εργασία και την παιδεία στα πανεπιστήμια ή στο σχολικό πλαίσιο. Τι διαφορές έχουν και τι ομοιότητες. Δεν θα σας μιλήσω για τη μεθοδολογία της μελέτης και που ακολουθήσαμε. Ε, μπορείτε να με ρωτήσετε στο τέλος. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η διτή εκπαίδευση που καλύπτει τις μαθητείες, την σχολική εκπαίδευση και την παιδεία γενικά, έχει δύο βασικές οδούς, δύο βασικά κανάλια εκπαίδευσης, τα σχολεία και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις βεβαίως δεν είναι μόνο παραγωγικές, αλλά είναι και τόποι μάθησης, ε, χώροι παιδείας. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ιδέα μίας ε, ε, ε, παιδείας εναλλαγής. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των χώρων εκπαίδευσης. Υπάρχουν διαρθρωτικές συνθήκες οι οποίες διαφέρουν ριζικά μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι φοιτητές οι μαθητευόμενοι ε, έχουν διαφορετικές συμβατικές υποχρεώσεις, διαφορετικό χρόνο εκπαίδευσης, διαφορετικούς ε, εκπαιδευτές ή δάσκαλους και αυτό που χαρακτηρίζει την μαθητεία είναι ακριβώς αυτή η διτή ειναι ακριβως αυτη η δυτη φυση της εκπαίδευσης. Τώρα πώς ε, διαμορφώνεται αυτή η διτή εκπαίδευση σχολείου μαθητείας είναι πολύ διαφορετική η τρόπη που εφαρμόζεται η υλοποίηση στην Ευρώπη. Τώρα το ερώτημα που θέσαμε, που θέσαμε είναι γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για αυτή την διτή ε, εκπαίδευση και να την υποστηρίζει. Τα τελευταία χρόνια διανύουμε μία μοναδική εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η παιδαγωγική έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί και πολλοί συμφωνούν ότι οι νέοι, οι νέοι αυτοί τρόποι μάθησης έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και έχει τεκμηριωθεί η αξία της πρακτικής μας Εγώ θα τονίσω ορισμένες πτυχές κλειδιά. Καταρχάς, ε, η μάθηση στον τόπο εργασίας μέσα στην επιχείρηση προσφέρει ένα αυθεντικό περιβάλλον, μια αυθεντική εμπειρία. Οι μαθητές έχουν αυθεντικές, πραγματικές σχέσεις, ζουν στην πραγματικότητα της επιχείρησης, ε, βλέπουν αμέσως το αποτέλεσμα της εργασίας τους και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σχολικό περιβάλλον που ε, ορισμένες φορές λειτουργεί σε στεγανό, δηλαδή δεν έχουν την άμεση επαφή με την πραγματικότητα και την εμπειρία η, εκπαίδευση, η μάθηση στον, ε, μέσω της εργασίας ή στον τόπο εργασίας προσφέρει την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, ε, επίσης αναπτύσσει μία επαγγελματική πλευρά του εκπαιδευόμενου του δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία στο το τι χρειάζεται για, μια για ένα επαγγελματικό προφίλ, χαρακτηριστικά, νοοτροπία, συμπεριφορές κλπ. Η οι ε, ε, έχουν, ε, προσφέρουν την ευκαιρία δημιουργίας ενός αξιόλογου εργατικού δυναμικού και σωστής εκπαίδευσης για τους νέους. Για να σας δώσω χαρακτηριστικά ποσοστά, στη Γερμανία 70% των μαθητευομένων βρίσκει δουλειά μετά από ένα μήνα, στην Φιλανδία 85% ανέργων νέων βρήκαν δουλειά μετά από μία περίοδο μαθητείας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά απασχόλησης μετά από μία περίοδο μαθητείας. Ε, ιδίως όταν μπορούμε να, να συντονίσουμε την ε, σχολική παιδεία με την ε, ε, επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχουν ε, βεβαίως ορισμένες προϋποθέσεις για μια επιτυχή μαθητεία και κατάρτιση. Οι εργοδότες πρέπει να επενδύσουν οικονομικά, αλλά το όφελος θα το δουν μετά από ένα χρόνο, διότι το όφελος προς τη θέμενη αξία θα είναι μεγαλύτερη από το κόστος το οποίο έχουν επενδύσει στον ε, μαθητευόμενο. Γενικά, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί σωστά στέρεα επιχειρήματα για την ενίσχυση των, της μαθητής και της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι όλες οι χώρες έχουν λίγο πολύ ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας. Αλλά το πώς ελκυστικά και προσφυλή είναι αυτά τα συστήματα, ε, εκεί έχουμε μεγάλη διαφορά αξιολόγησης. Δεν αξιολογούνται όλα τα προγράμματα αυτά το ίδιο. Δεν είναι όλα το ίδιο ελκυστικά. Πριν από δύο χρόνια έγινε μια μελέτη που έδειξε ότι 3,5 περίπου εκατομμύρια μαθητευόμενων υπήρχαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι περίπου το 1 τρίτο της επαγγελματικής κατάτησης, 3,5 ε, εκατομμύρια σε μαθητεία δηλαδή, μαθητευόμενοι και 5,5 εκατομμύρια σε άλλα προγράμματα εργασιακής ε, εκπαίδευσης. αυτό, αυτός ο προσανατολισμός της ε, επιχειρηματικής μαθητείας, αν θέλετε ακόμα, είναι στα σπάργανα. Μίλησα και για τα ωφέλη μιας τέτοιας εκπαίδευσης. Πάντα πρέπει να τα επενθυμίζουμε αυτά, αλλά εφόσον η μαθητεία είναι τόσο, τόσο καλή, έχει τόσα, τόσες θετικές πτυχές, γιατί δεν έχει ενσωματωθεί στα συστήματα παιδείας μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η τάση ενσωμάτωσης πολλών προγραμμάτων και ευρείας κλίμακας τέτοιας μαθητείας στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Καταρχάς, το ένα από τα βασικά ωφέλη είναι η απασχολησιμότητα και η δυνατότητα ε, ε, εξέβρεσης εργασίας σύντομα μετά τη μαθητεία. Ε, μπορεί σε ορισμένα παραδείγματα μάλιστα να έχουμε 100% επιτυχία ώστε κανένας να μην είναι άνεργος μετά από μία περίοδο μαθητείας. Όμως αυτό δεν είναι ακόμα κανόνας. Ε, υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Εκτός από τη Γερμανία, όλες οι χώρες που έχουν ε, συστήματα μαθητείας υπάρχει μία άνεση σχέση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ε, θέσεις τις οποίες ζητούν οι μαθητές για να εκπαιδευτούν, αλλά δεν υπάρχει η ισόβαθμη ε, δυνατότητα απασχόλησης. Υπάρχει λοιπόν μια ανισότητα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς. Και ένα άλλο θέμα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε είναι το ποσοστό εγκατάληψης από τα προγράμματα αυτά μαθητείας. Ορισμένα προγράμματα έχουν ένα υψηλό ποσοστό εγκατάληψης, 5% ε, και άνω σε ορισμένες χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, ε, 5% περίπου εγκαταλείπουν ε, το πρόγραμμα μαθητείας νωρίτερα από την ολοκλήρωσή του, που δεν σημαίνει πλήρη εγκατάληψη, αλλά γενικά ε, ας πούμε είναι πρόορη εγκατάλειψη ε, που πολλές φορές δεν οφείλεται, σε οφείλεται και σε προβλήματα που παρουσιάζουν οι μαθητευόμενοι στο χώρο εργασίας, ακαταλληλότητα κλπ η η μαθητεία είναι μία ε, δραστηριότητα, μία διαδικασία επιλογής. Είναι δύσκολο στην ηλικία 15-16 ετών να περάσεις μία επαγγελματική συνέντευξη, να επιλέξεις την κατάλληλη μαθητεία για σένα και είναι πολύ δύσκολο για τους νέους ανθρώπους που πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τον εαυτό τους ή τη γλωσσική ευχέρεια ή το θάρρος είναι λοιπόν δύσκολο σε αυτή την ηλικία. Δεύτερον υπάρχει και το θέμα των ε, διακρίσεων στην αγορά εργασίας και υπάρχει τάση να ε, προσλαμβάνει κάποιος πάντοτε έναν εργαζόμενο με το ίδιο προφίλ, με, με τις ίδιες προδιαγραφές. Και μια άλλη πρόκληση είναι η το, το, προχωρήσει κάποιος μαθητευόμενος στην περαιτέρω μάθηση, στην ανώτερη βαθμίδα πολλές φορές όταν ολοκληρώνουν ένα πρόγραμμα μαθητείας στα 17-18 μπορεί να έχουν ε, άλλες φιλοδοξίες, άλλα όνειρα. Το θέμα είναι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μια άλλη βαθμίδα, σε μια ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις της κατάστασης σήμερα και τώρα θα μιλήσω λίγο για το πώς ερμηνεύσαμε εμείς αυτήν την ε, ποικιλομορφία της εκπαίδευσης εναλλαγής. Υπάρχουν, όπως είπα, χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, που μπορούμε να πούμε έχουν ένα ολοκληρωμένο πλήρες πρόγραμμα, διτό πρόγραμμα ε, παιδείας. Ε, άλλες χώρες όπως ας πούμε η Γαλλία υπάρχει δυνατότητα μαθητείας ε, και επαγγελματικής κατάρτισης και συμβαδίζουν παράλληλα αυτά τα δύο και σε άλλες χώρες ε, υπάρχει, υπερέχει βεβαίως η σχολική παιδεία ε, και δεν μπορούμε να μιλάμε για, για μια σοβαρή επαγγελματική ταυτόχρονη κατάρτιση, μια δυνατότητα εναλλαγής και υπάρχουν ορισμένα στις χώρες, η Σλοβακία και η, η, η Τσεχία, ε, όπου η δυτή παιδεία ε, βασίζεται στο σχολείο. Δηλαδή γίνεται παράλληλα με τη σχολική εκπαίδευση. Στη Γερμανία, Αυστρία, και εκεί υπάρχει η παράλληλη εκπαίδευση μέσα στα σχολεία όπου υπάρχει η, σχολική παιδεία αλλά και η κατάρτιση. Άρα λοιπόν βλέπουμε πολλές διαφορές στα συστήματα. Όταν είπα ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη Γερμανία και την Αυστρία και Δανία, ε, τι περιλαμβάνει. Η μαθητεία αποτελεί έναν πολύ μεγάλο συντελεστή της όλης εκπαίδευσης. Η μαθητεία έχει ένα ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένο ε, και από πλευράς αγοράς εργασίας και από την πλευρά της παιδείας. Αποτελούν μέρη της επίσημης παιδείας και έχουν μία στενή διασύνδεση με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ένα πλήρες λοιπόν ρυθμιστικό πλαίσιο. Ποιες είναι τώρα οι προκλήσεις που παρουσιάζουν αυτά τα συστήματα. Ένα προφανές όφελος είναι ότι ε, παρουσιάζουν την δυνατότητα απασχόλησης και μελλοντικής εργασίας. Και σας είπα ότι τα ωφέλη είναι σημαντικά και είναι πολύ ελκυστικές αυτές οι δυνατότητες. Ορισμένα προγράμματα μάλιστα οργανώνονται από κοινού με ε, επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση όσον αφορά την, ε, την σύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή ε, όταν αποφυτούν είναι ενημερωμένοι στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και τα, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Και σε, αυτό το ολοκληρωμένο, σε αυτά τα ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουν αυτές ε, οι χώρες και η διαμόρφωση των προγραμμάτων είναι σαφής ε, και οι εκπαιδευτές είναι κατάλληλα ε, ε, καταρτισμένοι. Υπάρχει λοιπόν ένα σταθερό πλαίσιο και ευρεωμένο πλαίσιο. Όλη αυτή η προσπάθεια της διτής παιδείας εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την προθυμία εταιριών ή εργοδοτών να δεχθούν τους μαθητευόμενους ε, σε ορισμένες χώρες για τρία χρόνια. Ε, είναι λοιπόν μια πρόκληση, κατά πόσο είναι πρόθυμη και δεκτική. Ε, Πολλέ εταιρείε έχουν υψηλές και αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά το τι μπορούν να προσφέρουν στους μαθητευόμενους και ε, επειδή οι προδιαγραφές αυτές είναι αρκετά αυστηρές σε χώρες που έχουν ολοκληρωμένα προγράμματα, ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποθαρρύνονται και δεν θέλουν ή δεν έχουν το κίνητρο να εκπαιδεύσουν τους μαθητευόμενους. Και αυτό είναι λυπηρό διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές για την απορρόφηση των εργαζομένων, των νέων. Ένα, μία άλλη πρόκληση είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να προετοιμάσει τους μαθητευόμενους και να, ε, σε, σε, σε ε, την πλήρη εκπαίδευση, να τους προσφέρουν δηλαδή ένα πλήρες ε, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για, ώστε να μπορούν να επιλέξουν αργότερα διάφορες εργασίες ε, δηλαδή πόσες δεξιότητες μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αυτές ε, ώστε η αποφύτιση του, των μαθητευομένων να έχει μια συγκεκριμένη αξία. Και να μπορεί ο μαθητευόμενος όταν αποφυτεί να καλύψει όλες τις προδιαγραφές που χρειάζονται για την αγορά εργασίας. Τώρα, όταν η μαθητεία συμβαδίζει με άλλες μορφές εκπαίδευσης, η μαθητεία πολλές φορές δεν οδηγεί στις ίδιες, στα ίδια προσόντα τα οποία μπορούν να λάβει από διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης. Δεν είναι λοιπόν, είναι ένα ακόμα εμπόδιο, μία ακόμα πρόκληση πώς να διαμορφώνουμε σωστά τις μαθητείες αυτές ώστε τα προσόντα τους να αξιολογούνται ε, από την αγορά εργασίας. Και εδώ στο Βέλγιο ε, έχουμε γενικά ένα αρκετά σοβαρό ποσοστό εγκατάληψης της επίσημης ε, εκπαίδευσης και συνεχεία πηγαίνουν σε προγράμματα μαθητείας, περισσότερο σε παραδοσιακά σε παραδοσιακούς ε, τομείς. Και λιγότεροι μαθητευόμενοι πηγαίνουν στους τομείς υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας στην Ευρώπη. Στα προγράμματα που γίνονται παράλληλα με τη σχολική εκπαίδευση ε, δίνουν κάποια διπλώματα, κάποια πιστοποιητικά μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας, όπως στη Φιλανδία. Ε, και όπου η εκπαίδευση στην εργασία συμβαδίζει παράλληλα με το σχολείο, η μαθητεία σε μία επιχείρηση είναι πολύ πιο σύντομη. Δηλαδή, όταν η εναλλακτική μορφή ε, εκπαίδευσης ε, γίνεται μέσα σε μια επιχείρηση παράλληλα με το σχολείο, η περίοδος που μένει ο μαθητής στην επιχείρηση είναι πάρα πολύ σύντομη. Στη Γερμανία ε, υπάρχει μέσα στο σχολείο, δηλαδή ξεκινάει μια εκπαίδευση στην επιχείρηση, καταρχάς, η οποία συνεχεία αναπτύσσεται περισσότερο, ώστε στο τέλος της, του σχολείου να μπορεί κατευθείαν να μπει στην ε, επιχείρηση ο απόφυτος, ο τελειόφυτος. Υπάρχει επίσης και μια άλλη πρόκληση μεταξύ του τι μαθαίνει κάποιος σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση και τι μαθαίνει κάποιος στο σχολείο. Δηλαδή, αν είναι αξιόλογη ε, η μάθηση στην εταιρεία ή αν είναι πιο χρήσιμη η μάθηση στο σχολείο. Και εκεί καμιά φορά υπάρχουν αντικσότητες. Σας ε, παρουσίασε λοιπόν ορισμένες προκλήσεις, ορισμένα προβλήματα που υπάρχουν και οι συστάσεις τις οποίες καταλήξαμε λένε το εξής. πολλά, πολλοί φορείς που διαμορφώνουν πολιτική, εκπαιδευτική, η Κομισιόν, το Συμβούλιο Υπουργών, οι συστάσεις που εκδίδουν κλπ. Ελπίζουμε να λάβουν υπόψη τη διαφορά που υπάρξει μεταξύ χωρών όπως η Σλοβακία που δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε ένα σύστημα μαθητεία σε επιχειρήσει στα Σπάργανα, αλλά ένα πολύ καλό εξελιγμένο σχολικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουν σημασία στι διαφορές αυτές. Καλό είναι να ξεκινήσουμε από τη σχολική παιδεία και εν συνεχεία να ταυτοποιήσουμε ποιοι τομείς έχουν τις καλές δυνατότητες απασχόλησης και εξέλιξης και έχουν έλλειμμα εργατικού προσωπικού. Ε, πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τομείς όπου, όπου υπάρχει ζήτηση, ζήτηση απασχόλησης, ποιοι είναι οι τομείς ε, με οικονομική ανάπτυξη και να στοχεύσουμε συγκεκριμένα επιχειρήσεις, εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτά τα προγράμματα. Αλλά καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία και μέσα στο σχολικό σύστημα να δώσουμε τη δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης σε περιβάλλον εργασίας. Το σχολικό πρόγραμμα που ήδη περιλαμβάνει μια τέτοια πτυχή πρακτικής εκπαίδευσης θα πρέπει προοδευτικά και σιγά σιγά να αυξήσει το ποσοστό αυτό πρακτικής εκπαίδευσης, διότι είναι μία εξελικτική βαθμίδα, εξελικτική πορεία αυτή από το σχολείο, σιγά σιγά, στο εταιρικό περιβάλλον, συνεχεία στην απασχόληση στην εταιρεία ή στην εργασία γενικά. Όπου τώρα η μαθητεία γίνεται εκ παραλίλου με τη σχολική παιδεία, θα πρέπει αυτή η πρακτική παιδεία να οδηγεί σε συγκεκριμένα προσόντα, σε, μια, σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή διπλώματα. Πολλές φορές αυτά είναι άσχετα με τα ζητούμενα στην αγορά εργασίας και δεδομένου ότι η πρακτική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει ε, στην εκπαίδευση σε, σε, τομείς που έχουν ζήτηση και που ζητάν ε, εργαζόμενους, ζητούν εργαζόμενους, θα πρέπει τα πτυχία και αυτή η μάθηση που προσφέρεται να έχει ένα επίσημο πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν ε, επίσης να είναι ελκυστική, να προσελκύει νέους αυτή η πρακτική παιδεία, ιδίως ε, να βοηθήσουμε χώρες να καταρτήσουν την εκπαίδευση αυτή πιο ελκυστική, ώστε να, να την επιδιώκουν οι νέοι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξουμε την πτυχή της, ε, ε, του, την πολυ, πολυ, της, της της εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτει όλους τους νέους, όλους τους μαθητευόμενους, χωρίς διακρίσεις και να δίνει την ευκαιρία, να τους προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης. Αυτές είναι οι συστάσεις μας και σε άλλες χώρες αλλά, αλλά ειδικά στη χώρα μου τη Σλοβακία θα πρέπει να ξεκινήσουμε σχεδόν από το μηδέν ε, και άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα προχωρημένες. Εκεί καταλήξαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Λίτσνερ, και ευχαριστώ και την ομάδα σας η οποία επεξεργάστηκε ακριβώς αυτή την πολύ σημαντική μελέτη. Πιστεύω λοιπόν ότι πολλά από αυτά που ακούσαμε σήμερα καταδεικνύουν πόσο ζωτικός είναι αυτός ο χώρος. Έχουμε διασυνδέσεις που δημιουργούνται μεταξύ Υπουργών Απασχόλησης και Υπουργών Υπουργού Παιδείας. Η δυτή παιδεία λοιπόν προχωράει, προωθείται. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρήσιμο θα ήταν να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να επεξεργαζόμαστε ε, μελλοντικά με τον ε, νέο Επίτροπο. Και μεθοδολογικά είναι ενδιαφέρον, με την έννοια ότι η βάση είναι ευρεία όσον αφορά τις χώρες που έχουν υφιστάμενα συστήματα διτής παιδείας. Υπάρχουν υποδείγματα, μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται στην Ευρώπη που μπορούν να εμπνεύσουν τη μελλοντική μας εργασία. Εσείς εξετάσατε τομείς που υπήρξαν επιτυχείς και άλλοι ανεπιτυχείς. Επίσης είναι θέμα μεγέθους. Βεβαίως η Γερμανία έχει πολλές μεγάλες εταιρείες και μικρομεσαίες εταιρείες και συνεπώς μπορεί να βρει τα για να οργανώσει την δίτη παιδεία. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες ε, που έχουν μικρές επιχειρήσεις, για να μην πούμε και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οπότε όλα αυτά, αυτές οι χρηματοδοτήσεις ε, γίνονται πολύ δύσκολες. Άρα η προσέγγιση πρέπει να διαφέρει αναγκαστικά και ως προς το πρόγραμμα σπουδών αν θέλετε, υπάρχει μεγάλος συγκεντρωτισμός σε ορισμένες χώρες, σε άλλες χώρες υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τις διαδρομές σπουδών, ε, υπάρχει και η τεχνική εκπαίδευση ξεχωριστά. Όλοι οι άνθρωποι βεβαίως επιδιώκουν να ανέβουν, να προχωρήσουν στις ακαδημαϊκές ε, σπουδές τους και θα πρέπει να δημιουργήσουμε την ίδια περηφάνεια και για αυτούς που πηγαίνουν με απευθείας διαδρομή στην απασχόληση. Ερωτήσεις λοιπόν, η κυρία Καμαρέλα, που προέρχεται από μία από τις χώρες που αναφέρονται στην έκθεση. Ναι, ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης, ιδιαίτερα για τις συστάσεις σας ε, βέβαια δεν μπορεί κανείς ε, μέσα μια νύχτα να αναπτύξει ιδανικά συστήματα μαθητείας ε, και πρακτικής εκπαίδευσης χρειάζονται μεταβατικής περίοδο, μεταβατικές περίοδοι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σιγά σιγά βήμα βήμα και στη Γερμανία δεν είναι δεν έχουμε μόνο και αποκλειστικά διτή εκπαίδευση. Ε, πολλές φορές ε, οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι οι νέοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να απασχοληθούν, να αποσληφθούν και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να ε, μπορέσει και το σχολείο να προωθήσει τη μάθηση με συγκεκριμένα, και την απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων. Τα προσόντα ε, που θα αποκτήσουν είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ε, νέοι οι οποίοι δεν έχουν καμία εκπαίδευση πρέπει, πρέπει καταρχάς να μπουν στο σχολικό σύστημα και πριν από την αποφύτιση από το Λύκειο, ακόμα και στο γυμνάσιο, θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε σε αυτή την ηλικία να δούνε τον πραγματικό χώρο εργασίας, να γνωρίσουν πώς δουλεύει μια επιχείρηση και αν δεν το κάνουν αυτό ενδέχεται αργότερα να, έχουν, να με τόσο κακούς βαθμούς που κανένας δεν θα τους προσλαμβάνει. Εάν όμως έχει κάνει την πρακτική μαθητεία, έχει μια δυνατότητα, διότι μπορεί να πει ένας εργοδότης ότι μπορεί να είναι πάτος στα μαθηματικά ή στη, στα γερμανικά ή δεν ξέρω, σε κάποιο άλλο μάθημα, αλλά έχει κάνει πρακτική μαθητεία και έχει τα πρακτικά προσόντα. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα μοντέλα επειδή υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφορές. Στη Γερμανία είναι βασικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν. Αυτές προσφέρουν μαθητεία και εν συνεχεία οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι που ε, προσλαμβάνουν, αλλά την μαθητεία συνήθως την κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ πιο είναι, είναι υπέρμαχη μιας τέτοιας εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνη στην ε, προσφορά αυτών των προγραμμάτων μαθητείας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίω όσον αφορά χειρονακτικές ε, δεξιότητες, η εμπορική εκπαίδευση, οι εμπορικές ε, δραστηριότητες, αυτά είναι πάρα πολύ καλές και δεσμευμένες έναντι της μαθητείας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, ενισχύουμε και εμείς βεβαίως την ε, προσφορά μαθητείας. Είχαμε κάνει και μια εκστρατεία η οποία έλεγε όποιος δεν εκπαιδεύει πληρώνει. Δηλαδή, ε, δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο υποχρέωσης, συμβατικών υποχρεώσεων προσφοράς μαθητείας και για τις επιχειρήσεις αυτές. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τις πείσουμε, αλλά μερικές φορές πιάνει το σύστημα. Όχι ότι όλα είναι τέλεια στη Γερμανία, αλλά εντάξει. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας για τις ΜΜΕ. Η κυρία Τούμ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και η συνάδελφός μου ήδη ε, απάντησε σε ορισμένε από τις δικές μου ερωτήσεις, αλλά ήθελα και εγώ ε, να ρωτήσω πώς ε, μπορείτε να προσφέρετε κίνητρα σε αυτές τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τέτοια προγράμματα μαθητείας. Δεδομένου ότι μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι κίνητρα μπορούμε να προσφέρουμε όταν τους επιβάλλουμε, όταν τους ζητούμε να προσφέρουν μαθητείες πολλές φορές δεν υπάρχουν οι δυνατότητες μέσα στις επιχειρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν την ικανότητα ή τα χρήματα να προσφέρουν αυτές τις, ε, αυτά τα προγράμματα. Εγώ σκέφτομαι όχι τόσο πολύ τα σχολεία, αλλά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οι οποίες ε, φορολογούνται και πολλές φορές ε, δεν μπορούν να προσφέρουν. Πώς θα τους πείσετε, τι κίνητρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζάκανο τώρα. Δυστυχώς δεν έχουν μείνει πολλοί συμμετέχοντες στην αίθουσα, αλλά το θέμα είναι ζωτικό. Κρίσιμο. Ουσιαστικά μοιάζει σαν να πρόκειται να επινοήσουμε και πάλι τον τροχό. Ανάμεσα στους δύο πολέμους στη Ρουμανία είχαμε ένα τέλειο σύστημα το οποίο ακολουθούσε ακριβώς αυτές τις γραμμές. Δύο επίπεδα μαθητείας, ένα χαμηλό, ένα υψηλότερο. Από την ώρα που έφτανε στο υψηλότερο μπορούσε να φορέσει και καπέλο. Λοιπόν, μιλάμε πάλι για επαγγελματική αξιοπρέπεια. Δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε μηδενικά στη Ρουμανία και στη Σλοβακία. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζω λοιπόν να σας λέω ότι στη Ρουμανία οποτεδήποτε υπάρχει καυγάς σε πολιτικό επίπεδο κάποιος λέει αυτό μας είπε να κάνουμε οι Βρυξέλλες. Σαν να είναι άνθρωπος οι Βρυξέλλες που σου λέει κάτι να κάνεις. Όλοι επικαλούνται τις Βρυξέλλες και περνάει. Και γίνεται το πράγμα. Λοιπόν, εγώ όμως έχω πρόβλημα με αυτό πρέπει να σας πω. Αυτή η μελέτη Βεβαίως, θα την στείλω στον Υπουργό Παιδείας, αλλά θα ήθελα κάποιον από τις Βρυξέλλες να του, το στείλει, να του στείλει τη μελέτη, διότι ε, έρχεται, όταν έρχεται από τις Βρυξέλλες πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, κυρία Σούντροβα, με συγχωρείτε, είχατε ζητήσει για το λόγο προηγουμένως. Ναι, σύντομα κατά πάσα πιθανότητα ε, συμβαίνουν τα αντίθετα στη χώρα μας. Ό,τι προέρχεται από τις Βρυξέλλες υφίσταστε ε, αντίσταση. Ε, λοιπόν, αλλά και εγώ θα ήθελα η μελέτη αυτή να μεταφραστεί και να χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή απαρχή παρακολούθησης της κατάστασης, διότι αφορά κάποιες χώρες και ουσιαστικά θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και στα 28 κράτη-μέλη. Διότι αυτά είναι τα διάφορες εκφάνσεις μοντέλων που ακολουθούνται. Στην Τσεχία θέλουμε να σφυριλατήσουμε τη δυτή παιδεία και θέλουμε τελικά να μάθουμε τις βέλτιστες πρακτικές στις οποίες αναφέρεστε, ώστε να δούμε αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν για τη μελέτη και θα συνεχίσω να την παρακολουθώ. Πρόεδρος. Ο, κύστο, ο κύριος Μοργάνο τώρα, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η περίληψη αυτής της μελέτης θα μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες γερμανικά, αγγλικά ε, και γαλλικά θα έχετε την πλήρη έκθεση. Όπως αυτό συνηθίζεται. Κύριος Μοργάνο, ευχαριστώ πολύ για αυτή την θαυμάσια παρουσίαση και βεβαίως και για τη μελέτη. Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς που είναι πιο περίπλοκοι. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Πάρτε την Ιταλία. Το, η παιδεία υφίσταται αλλά υπάρχει μια διαφορά διότι η μαθητεία δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στη Γερμανία. Τεχνικό κολέγιο, τεχνική εκπαίδευση, εντάξει, αλλά έχουμε μια διαφορά. Έχετε τεχνική εκπαίδευση στο γυμνάσιο και μετά το γυμνάσιο επίσης και η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ιταλία σχετίζεται με το Υπουργείο Απασχόλησης και όχι το Υπουργείο Παιδείας. Να λοιπόν μια διαφορά όσο μας αφορά. Αλλά ολόκληρο αυτό το ζήτημα της μαθητείας μπορεί να ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις αν έχουν φορολογικά κίνητρα. Όμως, έχουμε μόνο μερική απορρόφηση αυτών των ρυθμίσεων ε, ανθρώπων οι οποίοι απασχολούνται μαζί, ενώ καταρτιζόμενοι. Γιατί το λέω αυτό τώρα, διότι κατά πάσα πιθανότητα αν ήμασταν σε θέση να επινοήσουμε κάτι πιο ομοιογενές, ένα σχέδιο πιο όμαλο, τότε θα μπορούσαμε να παρέχουμε κίνητρα τα οποία θα απέφευγαν τις μεγάλες διαφορές που βλέπουμε σήμερα μεταξύ κρατών. Και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί μία διακοπή όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Έχουμε τέσσερα λεπτά μόνο με τους διερμηνείς μας. Κάποιος είπε, και θα το υπογραμμίσω, ότι θα ήταν χρήσιμο αν είχαμε ένα κατάλογο από τις συντμήσεις που χρησιμοποιούνται. Αυτό θα μας βοηθούσε βεβαίως. Τα ακρονίμια δηλαδή. Ωραία. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες και σχετικές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω απαντώντας τις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μία αφορούσε το πώς, τι μπορεί να γίνει για να υποκινήσουμε τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το ζωτικό ερώτημα σε πάρα πολλέ χώρες, πρέπει να ομολογήσω. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχετε τα όσα μπορεί να κάνει το κράτος, φορολογικά κίνητρα δηλαδή, η εκπτωσή στην, ε, στις ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Στη Γερμανία υφίστανται για ορισμένου τύπους μαθητείας για τους νέους ειδικά που αντιμετωπίζουν δυσχερή κατάσταση. Αυτό είναι εφικτό στη Γερμανία γιατί υπάρχει το κεντρικό σύστημα καλά εγκατεστημένο και εγκαθιδρυμένο. Στις χώρες τώρα όπου η μαθητεία είναι κάτι καινούριο, υπάρχει ανάγκη ε, για την παροχή κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο ζωτικό ζήτημα πιστεύω ότι είναι ότι πρέπει να εξετάσετε πού εμφανίζονται οι ανάγκες. Ποιες είναι οι ανάγκες. Στην Εστονία όσον αφορά τις δεξιότητες ε, μπορεί να αφορούν τις υπηρεσίες και όχι την ε, βιομηχανία. Οπότε χρειάζεστε άλλου τύπου ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πρέπει δηλαδή να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα. Μπορεί να, χρειαζόμαστε, να μην χρειαζόμαστε κομμότριες αλλά λογιστές. Πρέπει πρώτα να εντοπίσετε τις ανάγκες στη χώρα σας και μετά θα βρείτε και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την απορρόφηση. Το δεύτερο που αναφέρθηκε ήταν η περιπλοκότητα της κυβερνητικής δομής, υπάρχει διχοτόμηση μεταξύ ε, των αρμοδιοτήτων. Ένα από τα βασικά στοιχεία που βοηθούν να προχωρήσουμε είναι η εγκαθίδρυση σαφών προτύπων προσόντων. Δηλαδή τι πρέπει στο τέλος του προγράμματος οι μαθητευόμενοι να έχουν μάθει, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερα ποιοτική ομοιογένεια στο πρόγραμμα και διασύνδεση μεταξύ σχολείου, σπουδών δηλαδή, και αγοράς εργασίας. Μελετήσαμε 10 χώρες, αλλά τις επιλέξαμε σαν αντιπροσωπευτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, λόγω των, συστημάτων τους επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίως ε, κοιτάξαμε και τα συγγράμματα ε, για πολλές άλλες χώρες. Κοιτάξαμε δηλαδή και τι έρευνα έχει γίνει σε άλλες χώρες. Θα δείτε λοιπόν ότι αναφερόμαστε συχνά στην Αυστρία, αν και η Αυστρία δεν περιλαμβανόταν σε βάθος ε, στη μελέτη. Τέλος, όσον αφορά την προθυμία για μαθητεία, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Όταν μιλάμε για μαθητείες, μιλάμε για νέους 15-16 ετών που πηγαίνουν στην επιχείρηση ε, και μια φορά που συζητούσαμε μία επικεφαλής ενός κέντρου ε, μαθητείας μου είπε ότι περιμένουμε να είναι όριμα τα παιδιά των 15 και 16 διότι ο εργοδότης θέλει ένα όριμο άτομο το οποίο θα συμβάλλει στην επιχείρησή του. Συνεπώς ως προς τις συμπεριφορές, τη στάση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι είναι έτοιμοι να κάνουν αυτή τη μετάβαση στην οριμότητα στα 15 και 16. Δεν είναι σύνηθες αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μήνες θα μιλήσουμε για αυτή τη ε, μελέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσία σας, για τη συνεισφορά σας. Νομίζω η μέρα αυτά είναι πολύ επικοδομητική, πολύ καρποφόρα. Θα τα ξαναπούμε στις 6 και τις 7 Οκτωβρίου. Γεια σας. Eh, ευχαριστούμε πολύ για τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε.